Okay. We are starting a little bit. Ξεκινάμε λοιπόν με λίγη καθυστέρηση μετά το μεσημεριανό. Θα συνεχίσω τώρα στα γερμανικά. Υπάρχει ένα γκολπ επισκεπτών από τη Γαλλία και τη Γερμανία που έλαβαν μέρος σε ένα διαγωνισμό που λέγεται πώς φαντάζομαι την Ευρώπη. Καλώς ορίζω αυτούς και τους συνοδούς τους. Χαίρομαι για το ότι υπάρχουν και Γερμανοί συναδελφοί, ο κύριος Κόλαν από την Πομερανία. Και ξεκινάμε από το επιπρόσθετο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την συνεδρίαση των συντονιστών οι οποίοι σήμερα τιμήθηκαν. τα όσα ορίζει ο νόμος για τη δική μας Επιτροπή και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων όσον αφορά τη νομική βάση του προγράμματος ε, πολίτη για την Ευρώπη. Εμείς θεωρούμε πως θα πρέπει να κινηθούμε στην ε, διαδικασία της συναπόφασης. Το τονίσαμε, ζητήσαμε από τους διάφορες, ε, ζητήσαμε από τις ομάδες μας, πλην του ECR και της GUE, καθώς η συνάδελφος σήμερα ήταν άρρωστη, ε, την άποψή τους και όλοι είπαν πως θα αρνηθούμε, θα απορρίψουμε αυτό το πρόγραμμα εάν δεν υπάρξει πρόοδος. Αλλά είμαστε διατεθειμένοι, αυτή ήταν τρίτη απόφαση που λάβαμε, να συνεχίσουμε στη διαδικασία της συναπόφασης. Θα συντάξουμε μια έκθεση. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την έκθεση, θα την υποβάλουμε σε Συμβούλιο και Κομισιόν και αναμένουμε Συμβούλιο και Κομισιόν να κάνουν έναν άτυπο τριμερή διάλογο μαζί μας. Εάν αυτός ο διάλογος δεν οδηγήσει στο αναμενόμενο αποτέλεσμα, σύμφωνα με ψηφοφορία των ομάδων μας θα απορρίψουμε το πρόγραμμα. Οπότε στείλαμε την προειδοποίηση, ελπίζω να ακούστηκε κάποιοι εδώ πέρα νεύουν, συγκατανεύουν, οπότε πήραν το μήνυμα πως είναι σοβαρό. Ακόμα δεν κάνουμε τίποτα, αλλά εάν δεν οδηγήσει πουθενά ο τριμερής διάλογος θα πούμε όχι. Το κατάλαβαν όλοι οπωσδήποτε οι εκπρόσωποι της Κομισιόν θα τα πούν αυτά στην Επίτροπο μαζί με τα χαιρετίσματά μας και βεβαίως ε, με το ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε ε, του προγράμματος αυτού. Ο Χάνου Τάκουλα είναι ο εισηγητής ε, και ε, βεβαίως ε, θα αρχίσει να ασχολείται με αυτό το θέμα γρήγορα. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα. Χαίρομαι για το ότι καλωσορίζουμε την Επίτροπο Εκπαίδευσης, Παιδείας, Πολυγλωσίας και Πολιτισμού, την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου. Έχουμε μιλήσει ήδη πολλές φορές, συχνά μεταξύ μας, παρουσία των εκπροσώπων, το ΣΥΝΣΚΙ και λοιπόν. Και βεβαίως για τα θέματα που μας απασχολούν το πρόγραμμα εκπαίδευση και νεολαία και το άλλο είναι το πρόγραμμα για τη δημιουργική Ευρώπη Γνωρίζετε πως δεν απορρίπτουμε τα πάντα, κάποια τα δεχόμαστε, πολύ περισσότερα από ό,τι πιστεύουν κάποιοι, αλλά βεβαίως έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και τα έχουμε πει ο κύριος Κορέλ ούτως ή άλλως είναι πάντα εδώ πέρα παρόν και τα σημειώνει φαντάζομαι και σας τα μεταφέρει τον... Ναι, ναι, στην επόμενη συνεδρίαση τον Ιούλιο λοιπόν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα και Σεπτέμβριο θα υποβάλουμε την έκθεση, το σχέδιο έκθεσης για το πρόγραμμα εκπαίδευση. Η κυρία Κώστα δεν είναι δυστυχώς εδώ πέρα αλλά και με αυτήν τα ίδια θα γίνουν υποβολή το Σεπτέμβριο. Εν ολίγης, λοιπόν, εν τω μεταξύ το Συμβούλιο επέτυχε μια κάποια συμφωνία για κάποιο περιεχόμενο του προγράμματος και νομίζω πως τώρα θα πρέπει να μας ενημερώσετε για το τι συνέβη στο Συμβούλιο και το τι γίνεται με τις ε, προτάσεις μας που είναι γνωστές. Χαιρόμαστε λοιπόν που είστε εδώ και αγαπητή Ανδρούλα έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, dear Doris, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Πέρασε αρκετό καιρό από την πρώτη μας συζήτηση για τα νέα προγράμματα και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνουμε έναν απολογισμό των όσων συνέβησαν αυτού τους μήνες. Θα ήθελα να αρχίσω ευθύ αμέσως με τα σχόλιά μου για το Εράσμους για όλους. Πιστεύω ότι στην Ευρώπη, η Ευρώπη σήμερα πολύ περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ένα ισχυρό και συνεπές πρόγραμμα που θα επενδύει ουσιαστικές ε, σημαντικούς πόρους στην παιδεία, στην κατάρτιση και στον αθλητισμό. Για κάθε ένα από αυτούς τους τομείς έχουμε θέσει σημαντικούς στόχους. Προτείνουμε να διπλασιαστούν οι ευκαιρίες για κινητικότητα και να δώσουμε μεγαλύτερες επιχορηγήσεις. Πάντοτε ε, ανταποκρινόμενοι στο κόστος ζωής στις διάφορες χώρες. Επίσης, για πρώτη φορά έχουμε ένα ευρωπαϊκό μέσο για τον αθλητισμό. Αλλά το πραγματικά ισχυρό σημείο του προγράμματος αυτού έγινε στη συνοχή του και στην αίσθηση σκοπού που το διαπνέει και νομίζω ότι όλοι εδώ θα συμφωνήσουμε και στις βασικές αρχές του. Πρώτα απ' όλα μια ε, σύγχρονη αρχιτεκτονική, ένα ενιαίο πρόγραμμα που θα μας επιτρέψει να καταρχήσουμε τους φραγμούς ανάμεσα στους διάφορους τομείς και να αναγνωρίσουμε ότι η τυπική και η άτυπη κατάρτιση δεν είναι δύο ξεχωριστοί κόσμοι. Αντίθετα αποτελούν ε, ε, μάλλον ε, κινούνται παράλληλα ο άτυπος με τον επίσημο τομέα, ενισχύοντας την προσωπική ανάπτυξη και προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση. Ένα ενιαίο πρόγραμμα καλύπτει αυτή τη συνέργεια. Δεύτερον, τρεις δράσεις, ένας πυρήνας τριών δράσεων που διατρέχουν ολόκληρο το πρόγραμμα και δίνουν ένα σαφές νόημα του τι έχει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυνατότητες μάθησης για τα άτομα, συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα όργανα για την καινοτομία και τις καλές πρακτικές και υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων των πολιτικών. Και τρίτον, μια σαφή σύνδεση ανάμεσα στις προτεραιότητες του προγράμματος και τους μακροχρόνιους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ισχυρότερο περισσότερο παρά ποτέ και δικαιολογεί τον προπολογισμό που έχουμε προτείνει. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι ακριβώς η καρδιά του προγράμματος Εράσμους για όλους και νομίζω ότι συμφωνούμε πάνω σε αυτά. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας, καθώς θα έρθουμε τώρα να εστιάσουμε σε θέματα για τα οποία γνωρίζω ότι έχετε ανησυχίες. Έτσι λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, συναντήθηκα με τους νέους πολλές φορές η τελευταία ήταν η σημερινή συνάντηση που είχαμε την νεολαία και που ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Αφιέρωσα χρόνο και άκουσα στις ανησυχίες τους σχετικά με το, τη συμμετοχή τους στο ενιαίο πρόγραμμα. Ε, συμμερίζομαι και σέβομαι τις ανησυχίες τους, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι βάσιμες. Ε, αν εμείς προτείνουμε να ε, υπάρχει μια σύνθεση της ε, ε τυπικής άτυπης ε, μάθησης και διαβίου προσέγγισης, το κάνουμε για να ενισχύσουμε τα συστατικά και όχι για να τα αποδυναμώσουμε. Οι ομάδες των νέων δεν θα χάσουν την ειδικότητά τους. Ε, αντίθετα, η δουλειά τους θα πάρει τη φυσική θέση που της ανήκει παράλληλα με όλες τις άλλες μορφές ανταλλαγών και συνεργασίας. Από την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη δημοκρατική συμμετοχή σε ανταλλαγές και στον εθελοντισμό. Οι δράσεις για την νεολαία θα αναπτυχθούν επίσης ώρες με, με τα υπόλοιπα τμήματα του προγράμματος και η κατάργηση των τεχνητών φραγμών ανάμεσα στους διάφορους τομείς της παιδείας και της κατάρτισης είναι ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα, ένα μήνυμα που το Κοινοβούλιο εδώ έχει ε, ε, διατρανώσει πολλές φορές. Είμαι σίγουρα υπέρ μια υψηλή ορατότητα τη νεολαία μέσα στο Εράσμου για όλου. Και είμαι πεπισμένη ότι αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσουμε ότι ο κλάδο αυτό θα ε, έχει όλα τα ε, ωφέλη ε, που ε, θα δίνει το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα και οι τρεις βασικές δράσεις. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το management. Το Erasmus για όλους θα εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο μέσω εθνικών φορέων. Ε, η εφαρμογή θα είναι και η υλοποίηση θα είναι πιο κοντά στους δικαιούχους από ό,τι είναι τώρα ε, και αυτό είναι κάτι που σίγουρα περιμένουν κάποιοι από τους επωφελούμενους. Αλλά εμείς θα έχουμε το καθήκον να εξασφαλίσουμε τη συνοχή και την αποδοτικότητα ως προς το κόστος. Γι' αυτό η Κομισιόν πρότεινε έναν ενιαίο φορέα συντονισμού, έναν ενιαίο οργανισμό συντονισμού για κάθε χώρα. Αλλά ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα ε, πάνω σε αυτό το θέμα, πιστεύω ότι παραμένει προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτύχει ε, μια πιο ομαλή και συνεκτική υλοποίηση του προγράμματος, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μέσα στο κάθε κράτος μέλος. Τώρα, για να έρθω στις δράσεις Ζαν Μονέ. Το γεγονός είναι ότι πολλοί νέοι θεσμοί θα μπορούσαν τώρα να ζητήσουν άμεση χρηματοδότηση από το Εράσμους για όλους. Όπως ε, οι έξι που αναφέρονται στο σημερινό πρόγραμμα ε, της διαβίου μάθησης το Κολέγιο της Πάρμας, παραδείγματο χάρη, το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και είμαι σίγουρη ότι ο καθένας από εσά ξέρει κάποια ε, νέα τέτοια εκπαιδευτικά ιδρύματα που ε, όλα περιμένουν, από ό,τι ξέρω, κάποια άμεση υποστήριξη από εμά. Αλλά κάθε διεύρυνση αυτού του καταλόγου των άμεσα εμποφελούμενων, αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε μια αντίστοιχη μείωση στον προϋπολογισμό που είναι διαθέσιμος για τους άλλους επιλέξιμους φορείς. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλους φορείς σε αυτόν τον κανονισμό. Ε, αντίθετα, θα έπρεπε να αφήσουμε όλους αυτούς τους φορείς να ανταγωνιστούν μεταξύ τους για χρηματοδότηση. Αυτή είναι η καλύτερη αγγίηση που έχουμε ότι θα υποστηρίξουμε τα καλύτερα project. Για τον αθλητισμό, απλώς θα ήθελα να καλωσορίσω την ευρύτερη συνένεση ε, σχετικά με το τι θα μπορούσε με χρήσιμο τρόπο να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα. Από κοινού ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ε, συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον αθλητισμό και επικροτώ την αφοσίωση αυτής εδώ της Επιτροπής σε αυτό το θέμα. Έρχομαι τώρα στις λεπτομέρειες της πρότασης έρασμος για όλους και του ελάχιστου προϋπολογισμού ανατομέα. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να σας δώσω περισσότερες εξηγήσεις και να σας προσφέρω και κάποιες ε, διαβεβαιώσεις για να σας καθησυχάσω. Προτείνουμε μια ευέλικτη νομική βάση η οποία θα επιτρέπει και θα ενθαρρύνει μάλιστα τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών κλάδων. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες δράσεις θα είναι ανοιχτές σε όλους τους κλάδους. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ακόμα μια φορά κάτι που είπα ήδη σε προηγούμενες ευκαιρίες. Οι κλάδοι, οι διάφοροι τομεί δεν θα πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι εξίσου ευπρόσδεκτοι, όποιο και είναι το μέγεθός τους. Δεν θα υπάρχει ε, μεροληπτική μεταχείριση υπέρ ε, ενός ή ε, του άλλου ε, τομέα. Στην ανακοίνωση που συνοδεύει τον κανονισμό προσδιορίζουμε τον ελάχιστο προϋπολογισμό που κάθε τομέας θα χρειαστεί για να πετύχει κάτι παραπάνω από τα ελάχιστα εγγυημένα από το τρέχον πρόγραμμα. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό, στην πρόταση της Κομισιόν κρατών κάθε τομέας θα λάβει ε, πολύ περισσότερη χρηματοδότηση από ό,τι συμβαίνει τώρα, σύμφωνα με προηγούμενη δέσμευση, δέσμευσή μας, ότι κάθε κλάδος θα υποφεληθεί από την αύξηση του προϋπολογισμού. Νομίζω λοιπόν ότι τα ερωτήματα που θα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι τα εξή. Είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε το 2012 σχετικά με τις λεπτομερείς προτεραιότητες της χρηματοδότησης, όχι μόνο για το 2014, αλλά επίση μέχρι το 2019 και το 2020 θα επιτύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ε, περικόπτοντας τον προϋπολογισμό σήμερα χωρίς να αφήσουμε, ε, μάλλον ε, προσδιορίζοντας την κατανομή του προϋπολογισμού σήμερα χωρίς να αφήνουμε καμία ευελιξία για το μέλλον ή θα πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να ανταποκριθούμε σε περισσότερα project που θα καλύπτουν διάφορου τομεί, κάτι που θα πρέπει να εθαρρυνθεί. Και τέλος θα ήθελα να σα πω δύο λόγια για το όνομα του προγράμματος. Περισσότερο από κάθε τι άλλο θέλαμε ένα όνομα που το, γενικό, το, το, το, πλατή κοινό αμέσω θα αναγνώριζε και θα δημιουργούσε ε, προσδοκίες σε αυτό. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν το πρόγραμμα Έρασμο σαν ένα από τα δέκα πιο επιτυχημένα και μεγαλύτερη ορατότητα ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όνομα αυτό έχει θετικά συνδεθεί με την εκπαίδευση, την κινητικότητα και τη διασυνορική συνεργασία ανάμεσα στα μυαλά εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Γι' αυτό, ε, κύριοι Ευρωβουλευτέ, ε, όταν θελήσαμε να προωθήσουμε την κινητικότητα στην επαγγελματική κατάρτιση, το Κοινοβούλιο ζήτησε ένα πρόγραμμα Έρασμο για του μαθητευόμενου. Και όταν θελήσαμε να αναβαθύνουμε την γνώση πάνω στην ε, πολιτική συνοχή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο ζήτησε ένα έρασμους για τους ε, ε, τοπικούς και περιφερειακούς ε, ερετούς εκπροσώπους. Και όταν θελήσαμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για, τους, για την κοινότητα των μαθητών, το ονομάσαμε Junior Erasmus. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε συνεπείς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δεν θα έπρεπε να απαρνηθεί την αρχή αυτή. Το ε, Εράσμους για όλους θα είναι πραγματικά για όλους. Θα προωθήσει την κινητικότητα όχι μόνο για τους ε, φοιτητές και τους μαθητές, αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση για τους ενήλικους και σε όλους τους τομείς και για την νεολαία. Και θα κάνει και πολύ περισσότερα πράγματα. Θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ της ε, παιδείας, της, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των οργανώσεων της νεολαίας. Θα προωθήσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και θα αναπτύξει τις καλές πολιτικές. Το Εράσμους για όλους θα στείλει ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους Ευρωπαίους που ασχολούνται με την ε, επίσημη, άτυπη και ε, τυπική ε, εκπαίδευση, ότι η Ευρώπη υπάρχει για όλους, ότι υπάρχει για να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και όλων των ε, δραστηριοτήτων των νέων. Και τέλος πρέπει να, αναρωτηθούμε το εξή. Τι θέλουμε περισσότερο από ένα όνομα. Θέλουμε έναν ορισμό ή ένα σήμα κατά τεθέν. Θέλουμε ε, μία φράση που να περιγράφει κάθε τι που κάνει ένα πρόγραμμα ή θέλουμε ένα όνομα που να απηχεί στους ανθρώπους και να συμβολίζει τις πιο, κάποιες από τις πιο βασικές αρχές της Ευρώπης. Την ευκαιρία, το ανοιχτό πνεύμα και τις ανταλλαγές. Επιτρέψτε μου τώρα σύντομα να έρθω στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και να αναλογιστούμε και πάλι τι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Πιστεύω ότι η πρότασή μας να έχουμε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την πραγματοποίηση του δυναμικού του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και για να προωθήσουμε την, το πολιτιστικό πλούτο και την ποικιλομορφία της Ευρώπης, αυτό είναι το εργαλείο που θέλουμε, ένα εργαλείο που θα ενισχύσει και την εγγενή αξία του πολιτισμού, αλλά και τον οικονομικό και κοινωνικό ρόλο του. χτίζουμε σε, σε, σε γερή βάση το Media ε, θα συνεχίσει την, ε, τις επιτυχείς δράσεις τους στην διανομή, την κατάρτιση και την δικτύωση για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο και μέσα και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κομμάτι του πολιτισμού θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους ε, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που αποφελούνται ήδη από το τρέχον πρόγραμμα. Αλλά δεν θα αποκλείσουμε ε, τους ε, οργανισμούς αυτό θα έστελνε λάθος μήνυμα προς τον ε, πολιτισμό και τους δημιουργικούς ε, κλάδους, αποθαρρύνοντάς τους από την αναζήτηση αναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Αυτό που είναι νέο στη δημιουργική Ευρώπη είναι η απόφασή μας να υποστηρίξουμε όλους αυτούς τους οργανισμούς με πιο αποτελεσματικούς τρόπους. Να γίνουμε για να γίνουν μάλλον πιο διεθνείς, να βρουν νέους εταίρους, να είναι καινοτόμοι και να αναπτύξουν και να ε, προσεγγίσουν νέα κροατήρια. Και εδώ θέλουμε μια πιο λεπτομερή νομική βάση. Αλλά και πάλι είναι ανάγκη να αναγνωρίσουμε ότι οι δημιουργικοί τομείς και ο κόσμος μέσα στον οποίο λειτουργούν αλλάζουν ραγδαία και σε βάθος. Η καινοτομία δεν μπορεί να προβλεφθεί και δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε λεπτομερώς που θα μας οδηγήσει κατά τη διάρκεια της 7 ετούς ζωής του προγράμματος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα στην νομική βάση. Το YouTube και το Facebook έχουν αλλάξει με ριζικό τρόπο τον ε, τρόπο με τον οποίο διανέμεται το οπτικοακουστικό περιεχόμενο και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό. Δεν υπήρχαν όταν σχεδιάσαμε το τρέχον πρόγραμμα Media και γι' αυτό προτείνουμε μια απλή, ευέλικτη νομική βάση που θα δίνει τη δυνατότητα προσαρμογών κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος. Όσον αφορά το μέσο εγγύσεων, η ε, μικρή και μεσαίοι οργανισμοί από όλους τους τομείς θα έχουν πρόσβαση στα δάνεια για τα οποία το μέσο αυτό θα εξασφαλίζει τις εγγύησεις. Συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων όσον αφορά το σχεδιασμό αυτού του μέσου και με χαρά μου μπορώ να σας πω ότι οι αρχικές δοκιμές ήταν αρκετά ενθαρρυντικές. Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω ένα σημείο το οποίο γνωρίζω ότι έχει δημιουργήσει ανησυχίες. Τα δάνεια δεν θα υποκαταστήσουν τις επιχορηγήσεις. Θα τις συμπληρώσουν. Ε, καλύπτοντας τις ε, ειδικέ επενδυτικές ανάγκες εκείνων των operators που έχουν την ικανότητα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Οι μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί θα συνεχίσουν να υποφελούνται από τις επιχορηγήσεις. Όπως είπα προηγουμένως, υποστηρίζουμε τον πολιτισμό και για την αγενή αξία του και για την οικονομική και ε, κοινωνική συνεισφορά του. Δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ εδώ μια φορά για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου για τα δύο αυτά προγράμματα. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαίο και ο πολιτισμός έχουν κρίσιμη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ε, σε ένα πνεύμα εταιρική σχέσης. Και με αυτό το πνεύμα είμαι ε, μαζί σας εδώ σήμερα και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας ε, για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει αυτή την εισαγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Μια που είμαι εισηγήτρια θα παραχωρήσω τον λόγο πρώτα απ' όλα στους συναδέλφους. Ξεκινάμε τη μαγιτέρη Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και εσάς κυρία Επίτροπε για την παρουσίαση αυτή που κάλυψε όλες τις πτυχές των προτάσεών σας. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση σχετικά με αυτή την πρόταση για τον ε, ενιαίο οργανισμό. Επαναλαμβάνω, για τον ενιαίο οργανισμό είναι η ερώτηση. Ε, πώς ε, μπορείτε να προβλέπετε στο μέλλον να επιβάλλετε σε ομοσπονδιακά κράτη ένα ενιαίο εθνικό οργανισμό. Δεν θα ήταν καλύτερα να κρατήσετε μια επιφύλαξη για να προβλέπετε μια ε, ρήτρα σχετική ε, ανάλογα με τη μορφή διακυβέρνηση ορισμένων ε, κρατών μελών. Γιατί φαίνεται ότι ο, ο ενιαίος αυτός ο οργανισμός είναι αντίθετο προ τα συστήματα ορισμένων ομοσπονδιακών κρατών όπου οι πολίτε είναι συνηθισμένοι σε κάποια μεγαλύτερη εγκύτητα που του βολεύει περισσότερο και που επιτρέπει και μια πιο απλή λειτουργία από ότι αν υπάρχει ένα ενιαίος εθνικό θεσμικός οργανισμός. Ε, θεωρείται ότι πρόκειται για μέτρο απλούστευσης ε, ε, ή, ή όχι, γιατί οι πολίτες που συναντούμε πάντοτε ζητούν μεγαλύτερη απλότητα σε κάθε διαδικασία ε, ε, στα πλαίσια όλων των προγραμμάτων. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας επ' αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Επίτροπε. Μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου. Ναι, ευχαριστώ που ήρθατε και για το ότι παρουσιάσατε το όνομα σας. Να αναφερθώ τώρα κάτι για, σε κάτι το οποίο είπατε. Μιλάτε συνεχώς για τους νέους. Όταν μιλάτε για τους νέους, Λοιπόν, να ξεκινήσω λοιπόν μιλώντα για του νέου. Κυρία Επίτροπε, λέτε πω ενδιαφέρεστε πολύ για του νέου. Τι όπως έχετε για την κατανομή ε, των κονδυλίων ειδικά για τους νέους. Δεν το ορίσατε αυτό και αντιλαμβάνεστε πως ε, στο Κοινοβούλιο δεν αρέσουν τα χαμηλά επίπεδα χρηματοδότησης που έχουν οριστεί εκεί γύρω στο 50%. Θα θέλαμε περισσότερα κονδύλια και θα θέλαμε να γνωρίζουμε και πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Και μιλώντας για νέους αναρωτιέμαι η πρότασή σας δεν αναφέρθηκε στην στήριξη των οργανώσεων νέων με διοικητικές επιχωρήσεις κτλ. μιλάτε για το φόρουμ αυτό της νεολαίας, αντιλαμβάνεστε πως είναι πάρα πολύ σημαντικές επιχορηγήσεις για τη λειτουργία αυτών των οργανισμών. Αρχικά βεβαίως μπορεί να φαίνεται πως ε, πολλές τέτοιες οργανώσεις ε, θα κλείσουν λόγω έλλειψης ε, οικονομικής στήριξης. Ξέρουμε πως είναι το πρόγραμμα για την νεολαία, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό νοτιούμε και το παρουσιάζεται ως ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να βοηθά την απασχόληση και την απασχολησιμότητα. Δεν είναι μόνο η απασχολησιμότητα το θέμα μας, είναι ο εθελοντισμός, ε, οι ενεργοί πολίτες ε, και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία αποτελούν μέρος του προγράμματος νεολαία σε δράση. Και μια και είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει και διαβίου μάθηση. Οπότε, πού βρίσκεται αυτή η πτυχή της ε, διαβίου μάθησης. Ε, π.χ. εθελοντισμός ε, ηλικιωμένων ή απασχόληση κτλ. Δεν ξέρω εάν είναι όλα αυτά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δεν θεωρώ πως είναι η πιο σημαντική συζήτηση αυτή, αλλά βεβαίως θέλω να πω κάποια πράγματα. Υπάρχουν ε, βουλευτές που δεν γνωρίζουν όλα τα προγράμματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Και όταν ζητάνε αυτοί οι βουλευτές να χρησιμοποιηθεί το Εράσμος για την επαγγελματική κατάρτιση ή για κάτι άλλο, μπορεί να μην γνωρίζουν το τι θέλει πραγματικά η Κομισιόν και το τι θέλει και η Επιτροπή που είναι επικεφαλής. Εδώ μιλάμε για Εράσμους. Αυτοί οι οποίοι υπέγραφαν το αίτημα αυτό δεν νομίζω πως ήξεραν ακριβώς περί την ασφαλή Δεν λέω πως είναι τέλειο το Εράσμους γιατί βεβαίως ήταν επιτυχές ε, και θα ήταν ε, και λανθασμένο να το υπονομεύσουμε. Υπάρχουν ε, και άλλα υποπρογράμματα που είναι σημαντικά και το σύστημα δανείων που υποστηρίζεται για μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμια. Χαίρομαι για το ότι μετά από μήνες συζητήσεων μάλλον ξέρουμε με τι θα μοιάζει, αλλά επίσης η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς θέλει και ποιοι είναι οι όροι θεωρώ πως ε, το Κοινοβούλιο δυσκολεύεται να συζητήσει πράγματα τα οποία δεν είναι εντελώς σαφή. Yeah, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε για αυτά τα οποία μας είπατε σήμερα. Ομολογώ ότι δεν χάνω ε, εύκολα την ψυχραιμία μου, αλλά αυτά τα οποία άκουσα σήμερα σχεδόν με έφτασαν σε αυτό το σημείο, γιατί βλέπω πως ε, έχουμε άλλο 1,5 χρόνο συζητήσεων. Δηλαδή, αν δούμε αυτά τα οποία μας είπατε και μεταξύ αυτών των οποίων ε, μας είχατε παρουσιάσει στην αρχή, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Είχαμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις όλοι μεταξύ μας, με τους συνεργάτες μας ε, και νομίζω πως είχαμε πάρα πολλές επιφυλάξεις, φόβους που εκφράστηκαν, πολλές ασάφειες όπου θέλουμε διευκρίνηση του προγράμματος. Νομίζω κατέστη σαφές ε, στη συζήτηση πως κανείς από εμά δεν είχε κανένα πρόβλημα με το streamlining και το πρόβλημα ε, να απλοποιηθεί το πρόγραμμα και να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση. Κανείς δεν είχε πρόβλημα με το να έχουμε ένα στιβαρό και συνεκτικό πρόγραμμα. Αλλά είναι σαφές τελικά πρέπει ο κόσμος να ξέρει ποια κομμάτια του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Και το πρόβλημα είναι, και νομίζω πως αυτό το έχουμε όλοι, πως μέσω του γεγονότους πως ε, τα ρίχνουμε όλα αυτά μέσα στο ίδιο τσουκάλι, πλέον σημαίνει πως κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να χρησιμοποιήσει από όλα αυτά. και το είχαμε και συζήτηση με τον κύριο Κορέλ, όπου η απάντηση ήταν «Μα είναι στο πρόγραμμα αυτά μέσα». Ε, ναι, αλλά όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι που επωφελήθηκαν από αυτό το πρόγραμμα και εργάστηκαν με αυτό το πρόγραμμα έχουν ακριβώς την ίδια εντύπωση με εμά, τότε ίσως και στην Κομισιόν πρέπει να τεθεί το ερώτημα μήπως δεν είμαστε Μήπω το πρόβλημα δεν είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να διαβάσουμε το πρόγραμμα, αλλά ότι αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μα είναι έτσι διατυπωμένο, ώστε, ε, να, μας ώστε να μην διαβάζεται και να μην μπορεί να μας καθησυχάσει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σωστή συνεργασία μαζί μας και θα ήθελα κάπου οι αμφιβολίες που εκφράζουμε εμείς και άλλοι να απαντηθούν και να πούμε ναι το τάδε σημείο πρέπει να το ξαναδουλέψουμε. Δεν φτάνει να λέμε πως ε, δεν θα, δεν θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους ε, μεγάλα και μικρά ιδρύματα. Ε, μα έτσι ξυπνάει ο φόβος πως θα υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλων πανεπιστημίων με άλλων ιδρυμάτων που εκπαιδεύουν νέους. Πρέπει λοιπόν να διατυπωθεί σωστά και ξεκάθαρα τι αντιστοιχεί σε ποιον, ποιοι στόχοι υπάρχουν στο κάθε κομμάτι του προγράμματος. Και θα ήθελα να εργαστούμε από κοινού τους ερχόμενους μήνες για να είναι ξεκάθαρο, συνεκτικό το πρόγραμμα έτσι ώστε πραγματικά να βοηθάει τον κόσμο και να μην ακούμε μόνο ως απάντηση «Α, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα» αν δεν το βρίσκει κανείς μέσα στο πρόγραμμα, δεν βοηθάει. Δεν, τι νόημα έχει, εντάξει, μπορεί να έχετε την ε, καλή θέληση. Αν δεν είναι γραμμένο κάπου, δεν μας βοηθάει τίποτα. Αυτή είναι η παράκλησή μου. Σας ευχαριστώ, φυσές. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, για τις εξηγήσεις σας. Να σας συγχαρώ για την πρόταση για αύξηση των προϋπολογισμών. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο κρίσης. Καταρχάς για το πρόγραμμα Jean ναι, θα ήθελα να εκφράσω την απορία μου. Εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με όργανα, με θεσμικά όργανα, τα οποία πρέπει να έχουν συγκεκριμένους στόχους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους και δεν θα πρέπει να υπάρχουν προγραμματισμοί οικονομικοί οι οποίοι να φύγουν τις μακροπρόθεσμες ε, ε, μορφές λειτουργίας τους. Απαιτούν οι οργανισμοί αυτοί μια κάποια δημοσιονομική ασφάλεια μέσα στην οποία να κινηθούν για να προγραμματίσουν σωστά τις εργασίες τους. Εδώ λοιπόν μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα. Και τώρα για το έρασμος για όλους. Όπως είπατε το έρασμος είναι κάτι το αναγνωρισμένο πλέον από όλους σχεδόν τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα Έρασμος έχει κάνει πολύ περισσότερα για την Ευρώπη από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Οι νέοι γνωρίζονται, μαθαίνουν γλώσσες, μορφώνονται και ταξιδεύουν. Και φοβάμαι λοιπόν ότι αν βαρύνουμε πολύ το πρόγραμμα Έρασμος θα το κάνουμε να χάσει λίγο την ταυτότητά του. Έχουμε άλλα τα Κομένιους, το Λεωνάρντο. Πώς θα ενταχθούν ουσιαστικά με τις προβλέψεις σας στο Έρασμος για όλους. Σαν παράδειγμα με το Έρασμος θα μπορούσα να πάω να σπουδάσω στην Ελλάδα, να συμπληρώσω τις σπουδές μου σε μια χώρα σαν την Ελλάδα αλλά με το νέο αυτό πρόγραμμα το οποίο θα είναι διαφορετικής φύσεως. Φοβάμαι ότι τέτοιου είδους αποφάσεις θα δυσκολευτούν. Ευχαριστώ e, πάρα πολύ για την παρουσίαση Έχω την αίσθηση ότι για το πρόγραμμα αυτό υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια λογική λύση, σε μια συμβιβαστική βέβαια λύση. Νομίζω ότι και με τη δική σας πρόταση μπορούμε να καταλήξουμε σε λύσεις οι οποίες θα καθησυχάσουν τους συναδέλφους που ανησυχούν. Στην ουσία αυτό το οποίο διακυβεύεται εδώ είναι η συνέχιση της χρηματοδότησης και κατά συνέπεια της λειτουργίας των προγραμμάτων για την νεότητα, ιδιαίτερα για κάποιες επιμέρους ε, κατηγορίες όπως ε, τις μη χαρακτηριστικές ή μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης. Νομίζω ότι τα προγράμματα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεχιστούν και στα πλαίσια του Εράσμος για όλους. Δεν θα πρέπει να απορροφηθούν και να χαθούν τα επιμέρους αυτά προγράμματα. Εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ υψηλό αριθμό ε, νέων που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προγράμματα και θα πρέπει να συνεχιστεί. Τώρα για τις ελαστικές δαπάνες. Είπαμε ότι για το έρασμος για όλους ένα κομμάτι θα είναι οι φοιτητέ και ένα άλλο κομμάτι θα είναι οι υπόλοιπες κατηγορίες των πολιτών. Αναρωτιέμαι αν το συνολικό ποσοστό, συνολικό ποσό, οι συνολικές πιστώσεις, πώς θα κατανεμηθούν, σε ποια ποσοστά θα καλύπτουν τη μία κατηγορία και ποια ποσοστά θα καλύπτουν την άλλη και γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία γύρω από τη λειτουργία όλων αυτών των επιμέρους προγραμμάτων. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τις πρωτοβουλίες σας, για την κατανομή των διαφόρων μέσων στον τομέα των κινηματογραφικών, σαν παράδειγμα στην ψηφιοποίηση. Και το πρόγραμμα Media λοιπόν έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει και καλύπτει ένα σημαντικό τομέα και θα καλύπτεται, καλύπτεται είμαστε βέβαιοι για τη λειτουργία του και για το 2013. Το πρόγραμμα Media έχουμε διαβεβαιώσει ότι θα συνεχιστεί εν πάση περιπτώσει στο μέλλον. Προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία το πρόγραμμα Media. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Κουρία. Ευχαριστώ Επίτροπε για τις συναντήσεις μας σε τόσο σημαντικά θέματα. Έχω την αίσθηση ότι η μορφή συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή είναι απαραίτητη για τη σωστή ε, κατάληξη των εργασιών μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ε, συμφωνήσουμε στα σημαντικά. Τι εννοώ. Εμείς ξεκινήσαμε από μία θέση σχετικά με το Erasmus for που προέβλεπε δύο διαφορετικά προγράμματα. Αυτό ε, το οποίο θα αφορούσε την νεότητα και αυτό που θα αφορούσε ε, γενικότερα τα θέματα εκπαίδευσης. Καταλάβαμε ότι το αίτημα αυτό ήταν κάτι ίσως το υπερβολικό, ήταν ίσως κάτι το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο, αν θέλετε, τη σωστή χρηματοδότηση των προγραμμάτων και γι' αυτό ακριβώς ε, δεχθήκαμε την ιδέα ενός ενιαίου προγράμματος. Αποδείξαμε, εν πάση περιπτώσει, την ευαισθησία μας και τη δεκτικότητά μας. Για τα θέματα της νεότητας όμως δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτά τα οποία λέγαμε πριν έξι μήνες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν το πρόγραμμα νεότητα θα έχει τη δική του ταυτότητα, αναγνωσιμότητα γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα περιπλέξουμε τον τρόπο λειτουργίας του. Και για το όνομα νομίζω ότι κανένας από εμά δεν θα πρέπει να επιμένει επί της αρχής το θέμα του ονόματος. Είναι ένα μέσο για να λειτουργήσει καλύτερα το πρόγραμμα και να γίνει καλύτερα γνωστό. Εσείς καταλήξατε στο Εράσμους για όλους. Εμείς τα συζητήσαμε αυτό, ακούσαμε απόψεις, ο καθένας έχει και διαφορετικές απόψεις ανάλογα και με τη χώρα του. Και πιστεύουμε ότι το Εράσμος για όλους ίσως να μην είναι το καλύτερο όνομα, αλλά σκεφτούμε κάτι άλλο εν πάση περιπτώσει. Ας μην είμαστε απόλυτοι. Εδώ μπορούμε από κοινού προς το συμφέρον όλων και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και φυσικά του Συμβουλίου θα μπορέσουμε να βρούμε ένα καλύτερο όνομα. Τώρα για, τις εθνικές, για τα εθνικά γραφεία, εσείς πιστεύατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο γραφείο αναχώρα. Από την άλλη είδαμε ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε διαφορετικές εμπειρίες οι οποίες είχαν ε, λειτουργήσει στο παρελθόν και έχουμε θετικές εμπειρίες. Από πλευρά σε πάση περιπτώσει, του Κοινοβουλίου σας διαβεβαιώ ότι προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανησυχίες τις οποίες έχετε εκφράσει και σε άλλα θέματα εσείς ε, ίσως όμως δείχνετε ότι εμένετε περισσότερο και δεν είστε διατεθειμένοι να μετακινηθείτε όσο εμείς θα θέλαμε. Ίσως λίγο μεγαλύτερη ευελιξία να ήταν χρησιμότερη. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, ήθελα να επανέλθω και εγώ στο θέμα του τίτλου του προγράμματος. Γιατί υπερασπιστήκατε το όνομα αυτό, ε, λέγοντας ότι είναι ένα brand το Erasmus και μια επιτυχής ιστορία. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ε, όσον αφορά την επιτυχία του Erasmus. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Όμως, ε, το επιχείρημα αυτό δεν θα μπορούσε να εξηγήσει τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ και μήνες. Γιατί και εδώ και έξω από το Κοινοβούλιο ε, πολλές NGOs και άλλοι οργανισμοί υποστηρίζουν ότι δεν είναι υπέρ αυτής της ονομασίας του προγράμματος και ότι βλέπουν πολλά προβλήματα μας λένε. Και αυτό είναι σημαντικό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Όχι να σκεφτούμε απλώς ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθος, είναι λίγο ανόητοι και δεν καταλαβαίνουν τη δικιά σας ιδέα σχετικά με αυτόν τον τίτλο. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε το όνομα του προγράμματος. Ήδη ε, εγώ έχω πει ότι υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι να το ονομάζουμε Education for All, γιατί καλύπτει και όλα τα προγράμματα εξ και δίνει ακριβώς το, το μήνυμα του τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτάσει σε όλους τους πολίτες της. Δεύτερον, ε, είπατε ότι η τυπική και η άτυπη εκπαίδευση δεν θα πρέπει να είναι κάτι που το βλέπουμε το ένα αντίθετο στο άλλο, ότι κάτι, δύο πράγματα που κινούνται ε, χέρι-χέρι. Ναι, αυτό είναι γεγονό από την άλλη μεριά υπάρχουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα και οι νέοι άνθρωποι έχουν ειδικέ κοινωνικές ανάγκες. Για να αντιμετωπιστούν αυτές είναι απολύτω κρίσιμη σημασία να έχουμε τις δυνατότητες αυτές για την μη τυπική, non-formal education, ε, γιατί διαφορετικά με την ε, επίσημη εκπαίδευση ε, προσεγγίζουμε μόνο ειδικέ κατηγορίες νέων. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ε, είναι σκόπιμο να διατηρήσουμε την προσφορά για non-formal education. Και η τελευταία μου παρατήρηση. Όπως και οι άλλοι, θα φαντάζεστε ότι είμαι και εγώ απολύτως υπέρ της ε, αύξησης του προγράμματος, ε, του, προϋπολογισμού για τη δημιουργική ε, Ευρώπη. Αλλά από το Συμβούλιο φαίνεται ότι η πρόθεση είναι να γίνει γενική περικοπή του προϋπολογισμού κατά 10% ε, παρόλο στις μεγάλες φιλοδοξίες που είχαμε για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το αποτρέψουμε, αλλά ε, δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα προβεί σε αυτές ε, τις περικοπές του προϋπολογισμού. Είναι, υπάρχει λοιπόν καμιά εγγύηση ότι το πολιτιστικό πρόγραμμα ε, δεν θα θυχτεί το Loans Facility, το μέσο εγγυήσεων για τα δάνεια δεν θα πειραχτεί ή ε, θα ε, γίνουν περικοπές και στα πολιτιστικά προγράμματα. Γιατί έκανα την ερώτηση αυτή στους συνεργάτες μου και μου είπαν ότι πρέπει να την απευθύνω σε εσάς διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν να μου απαντήσουν. Ευχαριστώ η κυρία Κώστα. Θα ήθελα να ασχοληθώ με το Δημιουργική Ευρώπη Ακούστηκαν γύρω από αυτό το πρόγραμμα αρκετές απόψεις με τις οποίες δεν διαφωνώ. Όπως είπε η κυρία Τρούπελ, είπε ότι θα πρέπει να τονώσουμε κάπως αυτή τη δραστηριότητα, αλλά μένοντας πάντα βέβαια στο πολύ χαμηλό αυτό ποσοστό του ΑΕΠ, δεν έχουμε πολλά δημοσιονομικά περιθώρια. Σχετικά τώρα με τις προτάσεις για τις νέες δημιουργικές τεχνολογικές και καινοτόμες δραστηριότητες και δημιουργίες, δεν είναι κακή ιδέα. Το σενάριο το οποίο αφορά τον πολιτισμό γενικότερα στα πλαίσια του ψηφιακού γενικά κόσμου είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει πάρα πολλές αλλαγές τα επόμενα δέκα χρόνια. Υπάρχουν ορισμένα θέματα όμως τα οποία χρήζουν εμβάθυνσης. Βλέπουμε σαν παράδειγμα ότι το Συμβούλιο Υπουργών στο ενδιάμεσο έγγραφό τους έχουν ε, εκφράσει κάποιες απορίες και κάνουν και ορισμένες προτάσεις οι οποίες θεωρώ ότι μας αφορούν σαν Επιτροπή Πολιτισμού. Και στα πλαίσια των συζητήσεων που είχαμε μαζί τους δείχνουν ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι ότι από τη μία δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε το νομικό πλαίσιο του Creative Europe, απ' την άλλη εγώ θα προτιμούσα εκτός από το, ε, να μην μπούμε για δημιουργική Ευρώπη, αλλά για πολιτιστική Ευρώπη, Cultural Europe καλύτερα και να έχουμε εγγυήσει ότι ε, το Μέντια θα συνεχίσει να έχει την δική του αυτόνομη ταυτότητα, να είναι πάντα αναγνωρίσιμο και να έχουμε την δυνατότητα να συνδυάσουμε τον πολιτισμό από τη μία και τις νέες αυτές ε, δημιουργικές ε, δραστηριότητες πολιτιστικές από την άλλη. Έχει υποθεί άλλωστε και από τα μέλη της Επιτροπής ότι μετά το 2014 το όνομα Μέντια, η ταυτότητα που έχει το Μέντια θα χαθεί και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ αρνητικό. Κοιτάξτε, ακούγονται πληροφορίες επίσημες και ανεπίσημες δεξιά και αριστερά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω λοιπόν τη διαβεβαίωσή σας σχετικά με την επιβίωση του ονόματος Μέντια. Στα πλαίσια τώρα του Creative Europe υπάρχουν ίσως κάποιες υπερβολικές πιέσεις για συγχωνεύσεις, οι οποίες μας κάνουν να χάνουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει ο πολιτισμός στον τομέα της αξιοποίησης της κοινή πολιτιστικής κληρονομιάς, ηλικής και άειλης, κάτι το οποίο δεν έχει, θα έλεγα, ε, τονιστεί αρκετά και αυτό το ξεχωρίζει από την βιομηχανική αν θέλετε διάσταση η οποία λειτουργεί σαν με κέρδος, με στόχο το κέρδος και στον τομέα πάντα τον πολιτιστικό και δημιουργικό. Λοιπόν, θα πρέπει αυτούς τους διαφορετικούς στόχους να τους σεβαστούμε και φυσικά να μην αγνοήσουμε και τον λεγόμενο τρίτο τομέα, ο οποίος εγκάρσια κατά κάποιο τρόπο καλύπτει και τους δύο προηγούμενους. Τώρα για το οικονομικό μέσο, το χρηματοδοτικό μάλλον καινοτόμο μέσο, αυτές οι ευρωπαϊκές εγγυήσει ε, για δανειοδοτήσεις είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε πρόωρο στάδιο. Ακούω τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Να θυμίσω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί σε διαφορετικές χώρες υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις. Σε ορισμένες χώρες τα θεσμικά ιδρύματα τα πολιτιστικά που χρηματοδοτούνται δεν μπορούν να ζητήσουν δάνεια Οπότε θα πρέπει εδώ να διασφαλίσουμε και για τα όργανα αυτά και για τις βιομηχανικές βέβαια και οικονομικές αυτόνομες μονάδες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να, δι, ε, να χρηματοδοτηθούν. Τώρα την τοπική διάσταση για την δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να τη δούμε αναπτυξιακά και όχι μόνο σαν μια δράση η οποία μπορεί να λειτουργήσει και σε διαμεθοριακό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να μην αγνοήσουμε την κοινωνική διάσταση του πολιτισμού. Ευχαριστώ κύριο Στάκουλα. Σύντομα παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Γεγονό είναι πως μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που ακούστηκαν είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσθέσουμε οτιδήποτε άλλο σε αυτές τις ε, ερωτήσεις. Η ερώτησή μου σχετίζεται με τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα μια ολοκληρωμένη άποψη. Ανισχούμε εδώ στην Επιτροπή μας για το πώς θα ε, ανταποκριθεί ο προϋπολογισμός σε όλες αυτές τις ε, προσθήκες Μιλάμε για προσθήκη 70%. Ελπίζω να το δεχτούν τα κράτη-μέλη και να μην περικόψουν τον προπολογισμό. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις ιδέες σας για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίτροπε, είμαι σίγουρη ότι θα βρεθούν ε, λύσεις ε, και στο ζήτημα του ονόματος και στο ζήτημα της αφήνειας των επιμέρους δράσεων στο πρόγραμμα προκειμένου να ε, αποφύγουμε τις ανησυχίες των ε, συναδέλφων για το ότι μπορεί να μην καλυφθούν δράσεις ή να πάψουν να χρηματοδοτούνται δράσεις που με την τρέχουσα με το τρέχον πρόγραμμα καλύπτονται. Ε, μπορούμε να σκεφτούμε προτάσεις για το όνομα, δεν έχω καμία αμφιβολία και είμαι σίγουρη ότι εσείς μπορείτε να το ξανασκεφτείτε, μιας και βλέπετε ότι η ολόκληρη Επιτροπή Πολιτισμού έχει τις αμφιβολίες της για το αν η αναγνωρισιμότητα αυτού του όρου θα ανταποκρίνεται στη σημασία και στη σκέψη που έχετε εσείς για αυτή την, ε, για την καινούργια έτσι, προσέγγιση αυτού του σύνθετου ζητήματος. Ε, εγώ δεν θα μιλήσω για τα επιμέρους ούτε το ενός ούτε το άλλου προγράμματος. Θέλω απλώς να σας μεταφέρω την αγωνία μου και ενδεχομένως να ζητήσω τη γνώμη σας για κάτι που μας απασχολεί εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και που δυστυχώς μοιάζει στα καινούργια προγράμματα που, που ε, βγαίνουν από την Κομισιόν και για την έρευνα, για παράδειγμα, που είναι εκτός της δικής σας ε, δικαιοδοσίας ε, ο πολιτισμός, αλλά με την ευρία έννοια του όρου, και είναι πάρα πολύ ευρία για να την ξεκαθαρίσουμε εδώ, συχνά είτε απορροφάται απευθεία από τα Υπουργεία Πολιτισμού των κρατών μελών, οπότε η, η, τα πανεπιστήμια να μην έχουν καμία δυνατότητα να διεκδικήσουν τέτοια προγράμματα. Και εδώ πρέπει να βρούμε μια λύση, πώς μπορεί ένα κομμάτι των προγραμμάτων του πολιτισμού να πηγαίνει στα πανεπιστήμια και όχι στα Υπουργεία Πολιτισμού μόνο και στις δράσεις τους, ένα. Και δεύτερον, πώς θα μπορούσατε, και εδώ θέλω απλώς να το σκεφτείτε, ε, να εντάξετε τη χρηματοδότηση των humanities μέσα στα προγράμματα της έρευνας. Κλείνω γιατί έχω μια απάντηση από, μια, από τη συνάδελφό σας την κυρία Κουίν σε μια ερώτηση που της έκανα για τον ορίζοντα 2020 όπου ε, το humanities νομίζω ότι κανένας δεν κατάλαβε ότι αφορά όχι τα human, αφορά τα humanistic studies και όχι τα humanitarian studies. Εδώ δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Παρακαλώ να μεταφέρετε την αγωνία των μελών αυτής της Επιτροπής ότι γίνεται ένα μπέρδεμα που στερεί κλάδους επιστημονικούς από οποιαδήποτε δυνατότητα χρηματοδότησης πέρα από τα πολύ λίγα που γνωρίζουμε σε ατομικό επίπεδο όπως είναι της, Madame, όπως είναι της Curie το πρόγραμμα. Ε, αυτά τα δύο κυρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο Βασιλείου για την παρουσίαση την οποία έκανε. Ε, δεν το είπαν άλλοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να το πω τουλάχιστον εγώ. Εμείς την πρόταση θα τη στηρίξουμε. Και θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο θέμα του ονόματος. Θα έχουμε συζητήσει όλοι οι, οι, οι ύποπτοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά συστηματικά θα έλεγα και ψάχνουμε να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις. Υπάρχει κάτι καλύτερο από την πρόταση η οποία έχει γίνει. Και το μόνο που έχω ακούσει είναι αυτό που είπε η κυρία Τρούπελ, που είπε ε, εκπαίδευση για όλους, education for all και όχι Erasmus for all. Είναι μια καλή εναλλακτική πρόταση. Ε, το συζήτησε το Συμβούλιο με την Προεδρία της Δανίας το θέμα αυτό. Δεν συμφωνούσαν όλοι ε, με το erasmus για όλους, αλλά απ' την άλλη δεν πρότεινε και κανείς κάτι άλλο. Οπότε αναρωτιέμαι μήπως μπορούμε ε, προσπαθώντας να βελτιώσουμε τα πράγματα να μην τα χειροτερεύσουμε παρακαλώ. Υπάρχουν ε, λοιπόν πάρα πολλά επιμέρους θέματα τα οποία τίθενται. Νομίζω ότι το Erasmus for All είναι αρκετά καλή πρόταση, αλλά αν ακούστουν και άλλες προτάσεις θα μπορέσουμε να τις εξετάσουμε και ίσως να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα ονόματα των επιμέρους προγραμμάτων σε μια δεύτερη βέβαια σειρά. Μπορούν να επιβιώσουν τα προγράμματα αυτά με το δικό τους όνομα. Απ' την άλλη εγώ τώρα την πρόταση της κυρίας Τρούπελ την οποία άκουσα και σημείωσα, τη βρίσκω ενδιαφέρουσα αλλά δεν είναι κάτι που θεωρώ καλύτερο από το Εράσμος για όλους. Τώρα τέρμα η συζήτηση για το όνομα. Έχουμε και τη διάσκεψη για τα 25 έτη του Εράσμου στην Κοπενχάγη και αναρωτιέμαι αν την ποιότητα του προγράμματος Εράσμους θα μπορούσαμε να την έχουμε μπροστά μας ε, ε, καλύτερο, με καλύτερο τρόπο. Ε, οι, οι μετακινήσεις Εράσμους χρήζουν περισσότερο εξέτασης. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία, όχι για το όνομα, την ουσία δεν αλλάζει με το όνομα. Το έχω εξηγήσει τόσες πολλές φορές που δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Το Εράσμος για όλους είναι ψέμα. Μα και το ε, Εράσμος ούτως ή άλλως, το κανονικό να λέμε Εράσμος ε, για όλους, δεν πάει γιατί μπορούσαν να πάνε μόνο όσοι έχουν λεφτά. Εράσμος σε άλλο τομέα, επίσης λάθος να το λέμε Τέλο δεν θέλω να εκνευρίζουμε, αλλά εκνευρίστηκα ήδη. Θέλω να πω ένα πράγμα μόνο. Κυρία Επίτροπε, σήμερα δεν μας είπε τίποτα διαφορετικό από αυτό που μας είπατε πριν από δύο μήνες. Όταν... Αυτά που μα έχει πει ο κύριο Κορέλ μία και δύο φορές, ο κύριος Μερές, τίποτα διαφορετικό. Ούτε ένα εκατοστό δεν υποχωρήσατε, παρά το ότι ξέρετε, και ο κύριο Κορέγια το ξέρει, το τι ακριβώς θέλουμε. Ούτε το τίτλο καν. Α, τέλος πάντων δεν είναι αυτό που θέμα σήμερα. Δηλαδή, έρχεστε εδώ πέρα και δεν μας δίνετε ούτε καν ένα σημάδι πώς λαμβάνετε υπόψη αυτά τα οποία λέμε. Και δεν μας λέτε τι ε, είπε το Συμβούλιο Επιδανικής Προεδρίας που έκανε μια δήλωση για το Ζαν Μονέ, έκανε μια δήλωση για την αποκεντρωμένη υπηρεσία, είπε πως είναι θέμα της χώρας της ιδίας και δεν μπορείτε να απαιτείτε από ένα ομοσπονδιακό κράτος, όπως είπε η Μαρή να τα κάνει όλα ένας. Προέρχομαι από τη Γερμανία. Δεν τα κάνει όλα ένας. Είναι θαυμάσια διαρθρωμένα τα πράγματα εκεί που υπάρχει και ο πελάτης. Δεν γίνεται να εξοδεύουν περισσότερα από ό,τι άλλοι στο ίδιο πρόγραμμα. Αυτό το οποίο κάνει η Μάλτα και το Λουξεμβούργο και οι άλλες οι μικρές χώρες. Δεν, δεν μπορείτε να, να μας αναγκάσετε χώρες οι οποίες δούλευαν μια χαρά να το αλλάξουμε, να το κάνουμε όπως οι άλλοι. Αφήστε κάποια επικουρικότητα εδώ πέρα. Και τι κάνετε. Μας λέτε, επιμένετε σε αυτά τα οποία υπήρχαν στο πρόγραμμά σας. Ε, είπατε πως θα υπάρξει κάποια διαφορά για ένα διαφορετικό πρόγραμμα για την νεολαία, αλλά πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο πρόγραμμα και να υπάρχει και μια γραμμή στον προπολογισμό. Και είπατε στον λόγο σας πολλές φορές ε, τη διαβίω εκπαίδευση. Δεν πρέπει. Ε, μάλλον σας αρέσει η έκφραση, το είπατε πολλές φορές. Εντάξει, καλός τίτλος. Μου ακούγεται, αλλά μπορεί να έχει και Helga δεν ξέρω. Λοιπόν, είπατε πώς θέλετε το θέμα Ζαν Μονέ και τα έξι ιδρύματα τα αμφισβητείτε. Μα δεν αμφισβητείτε έξι ιδρύματα. Τέσσερα αμφισβητείτε. Και δύο ρητό όχι. Δεν τα αμφισβητείτε. Και γνωρίζω πως αυτά τα δύο δεν τα αμφισβητείτε γιατί φοβάστε. Πως θα πει όλος ο κόσμος το ίδιο που λέμε και εμείς αν αμφισβητήσετε αυτά τα δύο. Πως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν είτε όλοι μέσα είτε όλοι έξω. και με αυτούς οι οποίοι θέλουν μέσα και την ε, Φλωρεντία και το άλλο ίδρυμα. Δεν γίνεται. Και την Πρίζ. Και αυτό είπε και το Συμβούλιο. Δεν είπατε τίποτα για τις προτάσεις του Συμβουλίου, άρα υποθέτω πως, άρα, πως και το Συμβούλιο είπε όλα μέσα. πως ε, πέριψε δηλαδή τις προτάσεις αυτές. Μετά είπατε πως θέλετε μόνο αυτό το, το μίνιμουμ ποσοστό. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε να είναι τόσο ε, ασαφές στο πρόγραμμα και να μην είναι δεσμευτικό. Εμείς θέλουμε να είναι δεσμευτικό. Και λέτε πως δεν ξέρουμε σήμερα τι θα γίνει το 2017 ή το 2019 και ποιες θα είναι οι απαιτήσει. Κοιτάξτε, ο χρόνος περνάει γρήγορα. Εμείς ξέρουμε το τι γίνεται και πόσα χρειαζόμαστε στον Λεωνάρδο. Χρειαζόμαστε περισσότερα από ό,τι χρειαζόμασταν τώρα. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ο Εράσμους. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ο Κομένιος. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Γι' αυτό θεωρούμε πως θα θέλαμε να ε, οριστεί το 80% του προγράμματος και μάλιστα εκεί που ανήκει κινητικότητα, συνεργασία, πολιτική έρευνα, αλλά μετά τα παρακαλώ σε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία σας το υπενθυμίζω είναι ονόματα και μάρκες. Δεν μπορεί να λέτε σε κάποιον ο οποίος εργάζεται σε αυτό το τομέα πως δεν ε, έχει πλέον σχέση με το Κομένιους. Οι άνθρωποι που ε, εργάζονται στο Κομένιους εδώ και χρόνια, 17 χρόνια, ε, έχουν σχηματίσει μια κοινότητα, ξέρουν τι είπα να πει Κομένιους. Επίσης το ίδιο και στα υπόλοιπα, Εράσμους, Λεωνάρδο κτλ θα βάλουμε αυτογκόλ εάν τα βάλουμε όλα κάτω από μια στέγη. Μπορούμε να διατηρήσουμε το όνομα, αλλά εντάξει μπορεί να έχετε δίκιο εδώ πέρα, να έχουμε μια προσέγγιση συνεργασίας, κινητικότητας, πολιτικής έρευνας, όλα αυτά μαζί. Εντάξει. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τα, τα πράγματα, να μπορεί ο καθένας να βρει το, το δρόμο του. Και Βεβαίω, η Κομισιόν, όσο και αν την εκτιμάμε, δεν μπορεί να έχει 44% χρημάτων να τα κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων, θα δώσουμε αυτό το 100 εκεί, αυτό το 100 εδώ και να μην... Εντάξει, έχετε και ανθρώπους ε, γνώστες ε, και νομικούς κτλ. λοιπά. Γιατί να ερχόμαστε και να λέμε Α, του χρόνου πρέπει να αλλάξουμε. Μα και να γίνει αυτό. Αν μα διαφωτίσετε βεβαίω, θα έρθετε, θα, θα μα ενημερώσετε και θα πούμε ναι. das gewählt ist. Νομίζω πως μπορούμε να ορίσουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε εμείς, οι οποίοι είμαστε και ιερετοί. Αυτό θέλουμε τόσο καιρό. Και ήταν εδώ πέρα οι συνεργάτες σας, και ε, είναι σε συνεχή επαφή μαζί μας. Και θα έπρεπε, ε, δεν ξέρω, να σας τα έχουν πει και αναμένουμε από εσά, αγαπητή κυρία Βασιλείου, κάποια μεγαλύτερη υποχώρηση, κάποια παραχώρηση προς τα εμάς. Πουθενά δεν μας έχετε παραχωρήσει ούτε ένα εκατεστό. Εντάξει, λέτε δεν έχουν υποβληθεί οι προτάσεις. Ναι, ε, τα, έχουμε πει όμως, τα έχουμε μιλήσει, θα υποβληθούν τον Ιούλιο. Και σας παρακαλώ μέχρι το Σεπτέμβριο να σκεφτείτε μήπως καλύτερα να αλλάξετε λίγο στάση. Και ναι, για το πρόγραμμα της νεολαίας. Καλά λέτε, θέλουμε άτυπη και επίσημη εκπαίδευση να είναι ισότιμες. Αλλά ε, ε, δεν θέλουμε να τα ανακατέψουμε. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την νεολαία και τις ενός νεολαίας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Το ότι ενδιάμεσα υπάρχει το Education and Youth και υπάρχει μια δυνατότητα συνεργασίας, ναι, αγαπητοί επίτροποι και αγαπητοί κομισιόν, μα αυτά τα λέμε πριν από πέντε χρόνια όταν δημιουργήσατε το lifelong learning. Ελπίζαμε, ελπίζαμε προς κάτω από αυτή την γενική στέγη θα μπορούσε να υπάρξει κάποια ανταλλαγή. Δυστυχώ δεν συνέβη. Εάν μπορέσει να συμβεί, θα χαρούμε ιδιαίτερα όσον αφορά τα λεφτά. Χαιρόμαστε για το ότι η Κομισιόν έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρό στην πρόταση, αλλά τι λάβαμε μετά. Δυστυχώ δεν ξέρουμε ούτε εμεί ούτε εσεί πρέπει να περιμένουμε να μιλήσει το Συμβουλίο. Και να πω κάτι ακόμα. Δεν ξέρω αν κατάλαβα σωστά ή αν παράκουσα και τα μάστερ, τα μεταπτυχιακά. Τα ζητάνε. Υπάρχει ζήτηση. να εγκριθεί κάτι το οποίο θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω ενός ταμείου εγγύσεων. Αλλά εάν δεν χρησιμοποιηθεί, γιατί τα ε, πρέπει να τα πληρώσει ο κόσμος ε, άμεσα ή αν τα πληρώσουν. Τι γίνεται, μένουν εκεί τα λεφτά, πάνε πίσω στους καθαρούς φορείς στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Τι γίνεται, θέλω να ξέρω τι θα γίνει με τα λεφτά γιατί είναι ε, λεφτά τα οποία κοιμούνται και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και θα χρειαστούμε ε, την εγγύηση το νωρίτερο του 2017, ίσως και το 2018, αλλά όχι πιο πριν. Και το, θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε τι θα γίνει εδώ πέρα και το ίδιο ισχύει και για τις δημιουργικές, το δημιουργικό κλάδο, ταινίε λοιπά. Αυτά ήθελα να ρωτήσω και άλλη μια ερώτηση. Οι κύριοι Κώστα και Βόρης και οι δύο αμφιβάλλουν για την συνέχιση του Μέντια. Σας παρακαλώ να μας διαβεβαιώσετε πώς θα συνεχιστεί. Ε, γιατί εμένα δεν με πιστεύουν. Ίσως πιστέψουν εσά. Ευχαριστώ. Shall we start with that? Yeah, please. It's yes. Easier. It's easier. Yes. Να αρχίσουμε με αυτό. Ναι, είναι εύκολο. Λοιπόν, ναι, θα συνεχίσει και θα ενισχυθεί το πρόγραμμα Media. Όχι με διαφορετικό πράγμα. Το brand media θα παραμείνει και το άλλο strand θα είναι ο πολιτισμός. Αυτό είναι σαφές. Μην κάνετε πράγματα που είναι ξεκάθαρα πιο πολύπλοκα. Θα ήθελα τώρα να επισημάνω ότι σε αυτή τη φάση δεν είμαστε ακόμα στη φάση των διαπραγματεύσεων. Σας παρακαλώ λοιπόν μην ανησυχείτε ότι δεν υποχωρώ στο α ή β σημείο. Γιατί σε κάποια φάση θα πρέπει να το κάνω. Θα πρέπει να το κάνω, αλλά πρέπει να ακούσω εσάς πρώτα. Άκουσα το Συμβούλιο και θα συνεχίσω να ακούω το Συμβούλιο και βεβαίως θα ακούσω και εσάς και σας έχω ακούσει πολύ προσεκτικά και σήμερα και την προηγούμενη φορά που ήρθα και βεβαίως κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε σε ποια σημεία μπορώ να υποχωρήσω εγώ και σε ποια σημεία μπορείτε εσείς. Ελπίζω ότι και οι δύο πλευρές θα κάνουν κάτι. Τώρα, ήθελα να πω ότι φαίνεται ότι τα πιο σημαντικά σημεία του Erasmus for All, το Erasmus για όλους, είναι πρώτα απ' όλα το όνομα η νεολαία και ο καταμερισμός των κονδυλίων και η Ζαν Μονέ. Λοιπόν, ας θα δούμε ένα-ένα. Να σας θυμίσω το εξής. Ο Έρασμος ήταν Ολλανδός, δεν ήταν Έλληνας. Δεν έχω λοιπόν κανένα λόγο να είμαι τόσο πολύ υπέρ του Εράσμου. Αλλά, ειλικρινά, όταν μιλάω με τον κόσμο, εγώ δεν ξέρω με ποιους μιλάτε εσείς, αλλά εγώ με όποιον μίλησα, όλοι το ξέρουν το πρόγραμμα Εράσμους. Το Εράσμους είναι το σύμβολο της κινητικότητας ο ίδιος ο έρασμος ήταν σύμβολο κινητικότητας. Ήταν κάποιος που πήγαινε από το ένα ε, πανεπιστήμιο στο άλλο. Μια εποχή που ταξίδευαν με κάρα ή με άλογα για να ε, εξαπλώσει ε, την ιδέα της κινητικότητας. Έτσι, αυτό το σύμβολο είναι ο έρασμος. Τώρα, αν σκεφτείτε ένα άλλο όνομα, η κυρία Τρούμπελ πρότεινε κάτι εναλλακτικό σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι σας έχετε κάτι κατά νου. Αν μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε μαζί με το Συμβούλιο ότι αυτό είναι καλύτερο όνομα από το Εράσμους, το θέμα είναι ότι εγώ θέλω ένα συνεπές όνομα. Ας το σκεφτούμε. Δεύτερο θέμα η νεολαία. Είπα στην εισαγωγή μου ότι θέλω η νεολαία να έχει μεγαλύτερη ορατότητα μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό δίνει κάποια μηνύματα. Στο τέλος θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό, αλλά στέλνει κάποια μηνύματα. Και γι' αυτό όταν μιλάω, μερικά πράγματα δεν μπορώ να τα πω πολύ ανοιχτά, αλλά χρησιμοποιώ πολύ προσεκτικά τις λέξεις για να δείξω τις προθέσεις μου. Έχετε απόλυτο δίκιο πάντως σε σχέση με τις ε, διοικητικές επιχορηγήσεις. Μετά από τις προτάσεις που ακούσαμε από την νεολαία, πριν καν διατυπώσουμε τη δική μας πρόταση, καταλήξαμε σε κάποιες δράσεις που θα είναι ένα πολυετές πρόγραμμα για τις οργανώσεις της νεολαίας που θα λαμβάνει υπόψη την πολυμορφία των δράσεων και το μακροχρόνιο των δράσεων. Δεν θα βασίζεται δηλαδή όλο αυτό σε ένα και μόνο project, αλλά σε ένα μακρόπνο πρόγραμμα. Και αυτό ε, ήταν ε, ε, ευπρόσδεκτο από τη μεριά τους. Σας λέω λοιπόν ότι κάποιες οργανώσεις της νεολαίας πρέπει να βασιστούν σε αυτές τις διοικητικές επιχορηγήσεις απλώς για να είναι σίγουροι ότι θα έχουν την γραμματιακή υποστήριξη που χρειάζονται για κάποια project. Τους λέω λοιπόν, ας συζητήσουμε, ας συνεχίσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτό. Και τους είπα χθε, υποβάλλετε τις δικές σας προτάσεις σχετικά με το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να διατυπώσουμε κάποια κριτήρια. Γιατί ειλικρινά δεν είμαι διατεθειμένη να δώσω διοικητικέ τέτοιε επιχορηγήσει σε 90 μη κυβερνητικέ οργανώσει, γιατί όλε ισχυρίζονται ότι κάνουν πανευρωπαϊκή δουλειά. Κάποιε είναι καταπληκτικέ οργανώσει, κάποιε άλλε όχι όμω. Και άλλαξαν οι συνθήκε σε σχέση με το παρελθόν. Τότε Είχαμε 15 κράτη-μέλη, τώρα έχουμε 28 και πρέπει να είναι ε, παρούσες και δραστήριες οι οργανώσεις αυτές σε πολύ περισσότερα κράτη-μέλη από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Σε 7 κράτη-μέλη έπρεπε να είναι εγκαταστημένες μέχρι τώρα. Αυτό δεν αρκεί πλέον. Καλό λοιπόν Κάλεσα τους νέους να υποβάλουν προτάσεις και κάλεσα επίσης και τις υπηρεσίες μου να συνεργαστούν στενά μαζί τους ώστε να δούμε πώς ε, μπορούμε τον καλύτερο τρόπο να εξυπηρετήσουμε αυτό το στόχο. Και εδώ συμφωνώ με την νεολαία, συμφωνώ με τους νέους ότι έχουμε ένα κοινό στόχο να εξυπηρετήσουμε εδώ. Γιατί η νεολαία είναι στο επίκεντρο όλη αυτής της προσπάθειας. Καταλαβαίνω ότι παραπονιέστε ότι δεν απαρίθμησα τι διάφορε δραστηριότητε που αφορούν τη νεολαία. Αλλά σίγουρα, αν αρχίσω να απαριθμώ όλε τι δράσει του προγράμματο Εράσμου για όλου, θα χρειαστούν πολύ περισσότερα από τα 15 λεπτά τη εισαγωγή μου. Θέλω όμω να επαναλάβω. Η εθελοντική δουλειά θα συνεχιστεί. Οι ανταλλαγέ νέων θα συνεχιστούν. Η κατάρτιση νέων εργαζομένων και η δικτύωση θα συνεχιστούν δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τιμάμε αυτή τη δουλειά, τη θεωρούμε αξιόλογη. Βεβαίως και τιμάμε την αξία της ε, ε, άτυπης και μη τυπικής ε, εκπαίδευσης και η πρόθεσή μας είναι να τις ενισχύσουμε και όχι να τις καταργήσουμε. Ο καταμερισμός του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι μπορεί να έχετε δίκιο από μία άποψη, ότι ίσως θα έπρεπε να αυξήσουμε τον καταμερισμό ανά τομέα, αλλά σίγουρα να αφήσουμε και κάποια ευελιξία. Θα ήθελα να σας μιλήσω για μια πραγματική εμπειρία μου. Μετά την ε, Αραβική Άνοιξη θέλαμε να κατανείμουμε κάποια κονδύλια για να προωθήσουμε μεγαλύτερη συνεργασία με τα πανεπιστήμια της Βόρειας Αφρικής. Και δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα λόγω έλλειψης ευελιξίας. Χρειάζεται να αφήσουμε λοιπόν ένα περιθώριο ευελιξία στα προγράμματά μας για να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε στις νέες συνθήκες, στις νέες ανάγκες ή με την ανεργία των νέων. Ένα μόνο συγκεκριμένο ποσό μπορούσαμε να αφιερώσουμε. βάσει των τοποθετήσεων του Εράσμους και του Λεωνάρντο λόγω της έλλειψης ευελιξίας. Ένα πολύ μικρό ποσό μπορέσαμε να αφιερώσουμε. Δεν είχαμε ευελιξία να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα κονδύλια. Τώρα, για το Ζαν Μονέ. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει η δουλειά των άλλων και επέλεξα μόνο τα δύο. Αλλά ε, χρειάστηκε να υιοθετήσουμε πολύ αυστηρά κριτήρια για να διατηρήσουμε την αριστεία. Και με δύο λόγια μόνο πραγματικά να σας πω ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, αυτής της μελέτης που πραγματοποιήσαμε ε, από έναν εξωτερικό οργανισμό αξιολόγησης για το Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης. Δεν δίνει επίσημα αναγνωρισμένα διπλώματα σε επίπεδο μάστερ ή διδακτορικού και δεν καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημών η Ακαδημία ε, Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, Δημόσιας Διοίκησης. Ε, εξαιρετικά ιδρύματα, αλλά παρέχουν χρόνια μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, εστιασμένα σε πολύ συγκεκριμένους τομείς το καθένα και πάλι δεν δίνουν επίσημα αναγνωρισμένα διπλώματα σε επίπεδο Μάστερς και PhD. Και τέλος, The European Agency κλπ. παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά δεν ασχολείται με ε, ακαδημαϊκά θέματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης που έγινε και κατέληξε μόνο στα δύο ιδρύματα, το Κολέγιο της Ευρώπης και στο, στην Προύζ και, στον άλλο, και το άλλο και ε, το Ινστιτούτο της ε, Φλωρεντίας. Όπως είπα όμως υπάρχουν και δεκάδες άλλα ιδρύματα που έχουν ε, ιδρυθεί έκτοτε που επίσης κάνουν πολύ καλή δουλειά και θα ήταν άδικο πιστεύω να το στερήσουμε αυτή την ευκαιρία. Γιατί καθένα, με κάθε ένα που προστίθεται στη λίστα θα μειώνεται το ποσό που πάει στο καθένα από αυτά τα ιδρύματα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι πιο δίκαιο να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό για όλα αυτά τα ιδρύματα και να δούμε κάθε φορά ποιο από αυτά πληρεί τις προϋποθέσεις. Τώρα για το πολιτιστικό πρόγραμμα. Μου κάνετε μια συγκεκριμένη ερώτηση και πολλοί υπουργοί μου έκαναν την ίδια αυτή ερώτηση όσον αφορά αυτό το μέσο ε, εγγύησης της δανειοδότησης. Αυτό το μέσο το θεωρούμε πάρα πολύ χρήσιμο και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πολύ τις πολιτιστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αν ο προϋπολογισμός μου περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορέσω να το καταφέρω αυτό το σημείο, θα προτιμήσω να το αφήσω απ' έξω και να μην θίξω καθόλου το πολιτιστικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα Media. Ήμουν σαφής, πάρα πολύ σαφής τώρα λέει η Πρόεδρος. Για το μάστερ, για τους φοιτητές, αυτό που έχουμε κατά νου είναι να αφιερώσουμε περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο για 55.000 φοιτητές το χρόνο. Αλλά βεβαίως, καθώς αρχίζουν να αποπληρώνονται τα δάνεια, θα μπορέσουμε να δώσουμε και άλλα δάνεια σε άλλους φοιτητές. Και πάλι θα επαναλάβω ότι αυτό δεν υποκοθιστά τις υποτροφίες ε, είναι συμπληρωματικό το μέσο αυτό ως προς τις υποτροφίες. Γιατί με ρωτάνε γιατί αντικαθιστάτε τις υποτροφίες ή τις επιχορηγήσεις από δάνεια. Ε, κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έχω τον προϋπολογισμό, να δίνω υποτροφίες σε φοιτητέ για να κάνουν μάστερ στο ε, εξωτερικό. Γιατί οι μελέτες μας δείχνουν ότι χρειαζόμαστε αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης, επίπεδο μάστερ δηλαδή. Πρέπει να το εθαρρύνουμε λοιπόν και να το υποστηρίξουμε. Αν είχα λοιπόν προϋπολογισμό να δώσω υποτροφίες για μάστερ θα το έκανα. Αλλά δεν το έχω. Μπορώ να δώσω μόνο σε ένα περιορισμένο αριθμό φοιτητών. Όμως αυτό το μέσο εγγύησης των δανείων πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει πολύ περισσότερους φοιτητές. Πρόεδρος, μπορώ να σας διακόψω. Αυτό σημαίνει ότι οι σπουδέ σε επίπεδο μάστερ ποτέ δεν θα πάρουν τι κανονικέ ε, υποτροφίες του Εράσμου. Όχι, σα λέω ότι δεν θα υποκαταστήσουν τα δάνεια τη υποτροφία του Εράσμου, πρόεδρο, γιατί υπόθηκε πολλέ φορέ ότι κανεί τώρα δεν θα μπορέσει να κάνει ανταλλαγή Εράσμου ε, για να κάνει μάστερ. Όχι, λέει η Επίτροπος, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορούν να πάρουν το Εράσμους αν θέλουν, αλλά θα είναι για έξι μήνες, ως συνήθως, αλλά το Master's Loan Guarantee θα είναι για όλη τη διάρκεια του Master, η δανειοδότηση δηλαδή, ε, για ένα-δύο χρόνια ανάλογα με τα μαθήματα που θα πρέπει κανείς να παρακολουθήσει. You, you, uh, στο ίδιο θέμα των... yes, please. I think, uh, Mrs. Νομίζω λοιπόν πως η κυρία Παλιαδέλη... Ε, μπορώ να με ακούσει τα ελληνικά. Σας το είπα ότι στο Marie Curie πρόγραμμα ενθαρρύνουμε, ενθαρρύνουμε τους φοιτητές, ε, όχι τους φοιτητές, τους, ε, ε, τους ερευνητές σε humanities να κάνουν αίτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές αιτήσει. Ίσως, και συμφωνώ εδώ, ίσως να χρειάζεται να δώσουμε περισσότερη δημοσιότητα στο γεγονός ότι το Marie Curie δεν ε, είναι για applied sciences αλλά και για τα humanities. Αυτά, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και θα πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή να οργανώσουμε διάφορες εκδηλώσεις που να δείχνουμε πραγματικά ότι τα humanities συμπεριλαμβάνονται σε αυτά. Τώρα, μου υποβάλλεται επίσης την ερώτηση γιατί να μην κάνουμε κάτι ούτως ώστε ε, τα grants να μην τα παίρνουν τα πανεπιστήμια, αλλά, ε, μάλλον όχι τα κράτη, αλλά τα πανεπιστήμια. Sorry. Ε, ναι. all cultural funds go to, to Συγγνώμη, μα όλα, όλα τα ταμεία αυτά, όλα τα, τα κονδύλια τα διαχειρίζονται τα Υπουργεία πολιτισμού. Οι δραστηριότητες πολιτισμού των πανεπιστημίων δεν επιτρέπεται άρα να συμπεριληφθούν. Ξεχωρίσω μεταξύ δύο πραγμάτων. Ό,τι δίδουμε εμείς από, το, ε, από τα δικά μας τα funds κάτω από το culture δεν πηγαίνουν στις κυβερνήσεις. Πηγαίνουν σε οργανισμούς. Και πάντοτε υπό τον όρο ότι αυτοί οι οργανισμοί συνεργάζονται με οργανισμούς άλλων χωρών. Ο λόγος είναι διότι θέλουμε να προωθήσουμε το cultural diversity, cultural cooperation, cultural dialogue. Ναι. Τώρα, εάν πάρουν structural funds, τα διαρθρωτικά ταμεία, για πολιτισμόν, τότε εκεί είναι τα κράτη. Και είναι τα κράτη-μέλη τα οποία ζητούν τι funds θέλουν να πάρουν κάτω από τα διαρθρωτικά ταμεία. Εμεί ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη. Και του λέω τώρα είναι, τώρα είναι η στιγμή που κάνουν τώρα τι συμφωνίε του με το DG Regio τι structural funds θα πάρουν και τους λέω να ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις μέσα στις συμφωνίες τους να έχουν και προγράμματα για πολιτισμό, για ε, infrastructure, ή κάτω από το Social Fund για training. Okay. Thank you very ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Επίτροπε. Άλλο ένα βήμα νομίζω κάναμε προς το νέο πρόγραμμα, όπως και αν λέγεται. Εγώ το ξέρω τώρα ως διαβίου μάθηση. Ε, είμαι ανοιχτή σε όλα πλην του Εράσμους για όλους. Λοιπόν, μπορούν όλοι να μιλήσουν. Έχουμε χρόνο μέχρι το φθινόπωρο και έχετε χρόνο στις διακοπές σας στην παραλία να σκεφτείτε ποιο είναι το καλύτερο. Και να σας πω κάτι κυρία Βασιλείου. Μίλησα με τους Κύπριους Υπουργούς και μου είπαν «Κυρία Πακ, ξέρετε στην Κύπρο, ο Έρασμος δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο Κομένιος. Οπότε χάρηκα για την νέα Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή επιτυχία στην Επιτροπή σας. Ε, κύριε Κορέλ, ε, συνεχίστε το έργο σας ε, σε επαφή μαζί μας. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Ωραία, περνάμε στην ανταλλαγή. Να πού πάνε όλοι. Έχουμε σήμερα καλέσει τον κύριο Κάλα και τον κύριο Πέτερς εκπρόσωπους ε, του Euronews. Ξέρετε πως από το 1993 έχουμε συνεργασία, η συγχρηματοδότηση του Euronews, με την Κομισιόν συγχρηματοδότηση του Euronews. Το Euronews λοιπόν δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να παρακολουθήσει κανείς σε 10 ευρωπαϊκές γλώσσες ε, την ευρωπαϊκή πολιτική. Αραβικά, τουρκικά, φαρσί, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ε, Ισπανικά και Πορτογαλικά. Γιατί γνωρίζουμε πως πρέπει να μεταδίδουμε και εκτός των συνόρων της Ευρώπης το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το κάνουμε εδώ και καιρό. Το κάνει δηλαδή το Euronews. Οι κύριοι που είναι εδώ πέρα σήμερα, Καλά και Πέτερς. Ο κύριος Πέτερς είναι πρόεδρος του Δουσού και ο Φιλιπ Κάλα ε, γνωστός μας. Είναι πρόεδρος της ε, της ανάπτυξης του Euronews. Ε, μας έχουν δώσει και ένα PowerPoint. 20 λεπτά θα έχετε και οι δύο. Ε, ό,τι πείτε σε αυτά. Μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε τι κάνετε βεβαίω με τα λεφτά μας. Γιατί ξέρετε πως υπάρχουν πολλοί που φθονούν ε, και αποφθαλμιούν ε, αυτά τα κονδύλια και θα πρέπει να είστε πιστικοί για να συνεχίσουμε να σας δίνουμε τα κονδύλια αυτά, τα οποία κατά την άποψή μου βεβαίως τα χρησιμοποίησατε σωστά. Εγώ είμαι ένας από τα 6,7 εκατομμύρια θεατές που βλέπουν μια φορά τη μέρα Euronews. Ό,τι γίνει μισή ώρα μετά το αργότερο το έχετε μεταδώσει. Κύριε Πέτρες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. το μέγεθος της παρουσίασης είναι αντίστοιχο με τη μεγάλη στήριξη που μας παρέχεται. Στην παρουσίαση την οποία θα κάνουμε, αυτό που έχει σημασία, πέρα από την εικόνα του Euronews που γνωρίζετε, να σας δώσουμε επιχειρήματα για το τι είναι το Euronews και τι απόσβεση των επενδύσεων σας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει κανείς από ένα τέτοιο κανάλι. Μεγαλώσαμε εδώ και 20 χρόνια που υπάρχουμε. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση περαιτέρω διεύρυνσης, μεγέθυνσης. Βλέπετε κάποιους αριθμούς στην πρώτη σελίδα. Σας δείχνουν ότι έχουμε 800 περίπου εργαζομένους, 25 διαφορετικές εθνικότητες, πολύ, λιγότεροι, ε, πολύ περισσότεροι συγγνώμη, από τους 200 που υπήρχαν στο παρελθόν, χάρη στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε και 100 νέους υπαλλήλου, γιατί θα ξεκινήσουμε με τα ελληνικά και τα ουγγρικά παρακαλώ στο Euronews. Έχουμε τη στήριξη 20 μετόχων δημοσίων ε, σταθμών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ικανοί σήμερα μέσα από τις 11 γλωσσικές μας υπηρεσίες να απευθυνθόμαστε σε 3,5 ε, δις, εκατομμύ... σε δις πολίτες του κόσμου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την παγκόσμια αγορά. Έχουμε μια πολιτική πολύ σημαντική διεύρυνση στα τελευταία δύο χρόνια. Περάσαμε από δύο εξωτερικά γραφεία σε 14 με το ανοίγμα δύο γραφείων στην Αθήνα και στη Βουδαπέστη. Ανοίξαμε επίσης και ένα σημαντικό γραφείο στις Βεξέλλες, το πιο σημαντικό διεθνές χάρη στη στήριξη της Ένωσης και όπως βλέπετε στον πίνακα αυτό τώρα είμαστε παρόντες στη Ουάσιγκτον, στην Τόχα, στο Ντουμπάι, τον Αύγουστο θα ανοίξουμε μάλλον στη Washington και ανοίγουμε όλο και περισσότερα γραφεία ανταποκριτών στον υπόλοιπο κόσμο. Για την Αθήνα και τη Βουδαπέστη θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε δύο γλωσσικές ε, μορφές του καναλιού μας με τοπικό τρόπο. Όχι ε, συγκεντρωμένα όλα στη Λιόν, αλλά από υπηρεσίες επιτόπου στην Αθήνα. Θα υπάρξουν 30-35 άτομα και άλλα 30-35 άτομα στη Βουδαπέστη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη πρεμιέρα για το Euronews και νομίζουμε ότι το σύστημα αυτό είναι χρήσιμο. Ε, θα ξεκινήσουμε εκτός από τα ελληνικά και τα ουγγρικά. Ε, είχαμε ξεκινήσει άλλες πέντε γλώσσες μη ευρωπαϊκές τα τελευταία χρόνια. Δεν επιμένω πάρα πολύ σε αυτά, ίσως να υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις. Το Euronews όπως και κάθε τηλεοπτικό σταθμός δεν θα πρέπει να είναι ένας απλός τηλεοπτικός σταθμός, αλλά σαν μια μεγάλη θα έλεγα πλατφόρμα η οποία θα καλύπτει με την παρουσία του τις ανάγκες ε, της κίνησης, σαν παράδειγμα ε, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, σταθμοί. Έχουμε υπογράψει πάρα πολλές συμφωνίες επίσης με τους κατασκευαστές τηλεοράσεων καλύπτουμε το 93% των παραγωγών σε σχέση με την λεγόμενη συνδεδεμένη τηλεόραση. Ξέρετε ότι αγοράζετε σήμερα μια τηλεόραση, το βάζετε στο διαδίκτυο και για να είστε παρόν θα πρέπει να αναπτύξετε applications όπως ακριβώς γίνεται για τα iPhone. Και ε, καλύπτουμε με την παρουσία μας το, 95, το 93% των τηλεοράσεων, των νέων τηλεοράσεων. Ε, είμαστε επίσης και στον τομέα των κινητών τηλεφώνων παρόντες και επίσης στα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα. Κάτι το οποίο είναι λογικό για με ένα κανάλι πληροφόρησης όπως το δικό μας. Όπως βλέπετε το 1993 ήμασταν 18, σήμερα είμαστε 200 αυτό δεν διευκολύνει, εν πάση περιπτώσει, ενώ το αριθμός των καναλιών ε, είναι 200 σήμερα. Ε, το Eurosport έχει ένα κάποιο μονοπόλιο γιατί δεν υπάρχουν άλλα αθλητικά διεθνή κανάλια. Για μας όμως ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός. Παρ' όλα αυτά έχουμε πλέον εκτήματα απέναντι στους ανταγωνιστές μας Προσπαθούμε εμείς να αντισταθμίσουμε την αμερικανική αντίληψη για την ενημέρωση και το έχουμε πετύχει. Γιατί στην Ευρώπη μας βλέπουν σήμερα καθημερινά 5,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Αριθμοί όχι πολύ γνωστοί, αλλά άμα δείτε με το CNN και το BBC News που δεν ξεπερνούν το ένα τις 200.000 και το άλλο κάτι παραπάνω από ένα εκατομμύριο βλέπετε ότι προχωράμε καλά. Η κριτική είναι ότι το Euronews χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε εδώ λίγο. Η κατανομή των εσόδων του 2011 δείχνει ότι υπάρχει μια ισορροπημένη στήριξη από τους μετόχους οι οποίοι χρηματοδοτούν το κόστος των αδειών για να χρησιμοποιούν το κανάλι μας σε διάφορες γλώσσες, πορτογαλικά, ρωσικά, τουρκικά τα δικαιώματα λοιπόν, και αυτό είναι το 30% των εσόδων μας, οι μέτοχοι, και 30% παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επανέλθω σε αυτά προηγουμένως, και ε, έχουμε 40% εμπορικά έσοδα. Τα περισσότερα από τα έσοδα αυτά τα επενδύουμε στην σύνταξη του καναλιού γιατί είναι ένα 37% του κόστους λειτουργίας της ε, Euronews και φυσικά έχουμε και το τεχνικό κομμάτι που απορροφά το 26% των εσόδων. Θα μπορούσα να σας πω ότι το Euronews είναι ο πιο ωραίος και πιο καλός σταθμός στον κόσμο. Για να σας πείσω θα πρέπει να μιλήσουν οι άλλοι για μας. Και θα σας παρουσιάσω μια αξιολόγηση την οποία ζήτησε να γίνει το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ανανέωσε το, στη σύμβαση πλαίσιο από μια εξωτερική υπηρεσία και υπήρξε μια έκθεση αξιολόγησης 250 σελίδες. Το πρώτο κομμάτι λέει ότι αυτή η υπηρεσία αξιολόγησης λέγει ότι το Euronews ανταποκρίνεται στις στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το Euronews σήμερα είναι ικανό να γίνεται κατανοητό θα έλεγα από τους ακροατές του, τους τηλεθεατές που δεν είναι πολύ ενημερωμένοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις λεπτομέρειες. Και γι' αυτό το, New, το Euronews είναι μια μορφή εκλαΐκευσης των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ταυτόχρονα λέγεται ότι το Euronews θα μπορούσε να διεκδικήσει αν θέλετε, την παροχή μιας πραγματικά ευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας και να διαμορφώσει ένα νέο ευρωπαϊκό κενό, κοινό, συγγνώμη. Δεν έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα βέβαια των, των καναλιών των εθνικών, δεν είμαστε μάσκαριες, και νομίζω ότι αυτοί μπορούν να μεταφέρουν εμάς ενώ εμείς δεν μπορούμε να τους μεταφέρουμε αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολυνθούν κάπως τα πράγματα αυτά. Δημιουργούνται κάποιες εθνικές ε, μορφές ε, καναλιών ενημέρωσης και χρησιμοποιούν νέα δίκτυα διανομής, κάτι το οποίο είναι ένας επιπλέον ανταγωνισμός. Λέγεται πάντα σε ε, σε αυτήν την έκθεση της υπηρεσίας αξιολόγησης ότι το, οι τιμές τις οποίες προτείνει το Euronews είναι ανταγωνιστικές, συγκρίνουν και κάποια άλλα προγράμματα που πολλούσαν άλλες εταιρείες σε άλλες γενικές διευθύνσεις και είπαν ότι είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί. Δεν πληρώνεται πιο ακριβά λοιπόν για το Euronews αυτά που πληρώνεται ακριβότερα αλλού. Υπάρχει ένας αριθμός πολύ ενδιαφέρον εδώ την Adventia το 2009 600 λεπτά ανεβδομάδα για ευρωπαϊκά θέματα, ενώ το BBC World και το Deutsche Welle που αξιολογήθηκαν επίσης δεν αναφέρονται παρά μόνο 10 ε, φορές λιγότερο στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είμαστε σχεδόν στα 1500 λεπτά την εβδομάδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Βλέπετε ότι από το 2009 μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να ανοιγόμαστε όλο και περισσότερο στα ευρωπαϊκά θέματα. Δεν μπορώ να κάνω μια παρουσίαση στο ευαγέ σας ίδρυμα αν δεν αναφερθώ ακριβώς ε, στη συνεργασία μας με τους ευρωβουλευτές που έχουν σημαντικό ρόλο ε, στο κανάλι μας. Εδώ είναι κάποιες από τις τελευταίες παρεμβάσεις ε, των Ευρωβουλευτών στο Euronews. Δεν φτάσαμε στα μέλη της Επιτροπής σας, δεν σταθήκαμε τόσο πονηροί. Αλλά βλέπετε ότι κάθε φορά που υπάρχει κάποιο σημαντικό θέμα για συζήτηση απευθύνουμε, ε, θα έλεγα συστηματικά, απευθυνόμαθα συστηματικά στους Ευρωβουλευτές ε, οι οποίοι θεωρούμε ότι εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα να επιμείνω σε ένα κομμάτι αρκετά σημαντικό να πω ότι τέλει δεν είμαστε, μπορούμε να βελτιωθούμε. Πάρα πολλοί θεωρούν επίσης ότι ο ρόλος του Euronews δεν έχει πλέον, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί πλήρως και ότι μπορεί να πάει και πολύ καλύτερα. Κοιτάξτε, αυτό ε, μπορώ να σας το πω ότι πράγματι έχουμε δυσκολίες σαν κανάλι να μιλήσουμε για την Ευρώπη σήμερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Είστε οι πρώτοι που θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι δύσκολο για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα αυτά και να τα συζητήσει ε, στα κανάλια. Έχουμε πολλές προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι πρέπει να απευθυνθούμε και σε τοπικό κοινό αλλά και σε ευρωπαϊκό κοινό. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προσδοκίες από τα μέσα ενημέρωσης. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μετασχηματίσουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε πηγές και να τα όλα αυτά σε ειδήσει ενδιαφέρουσες, ξέρετε, σαν παράδειγμα με τις συναντήσεις κορυφής. Όταν έχουμε την, την τύχη βέβαια να κυνηγάμε τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη που μιλάει στο τηλέφωνο του επί 3,5 ώρες, έχουμε εικόνες, αλλά αλλιώς οι εικόνες δεν δείχνουν τρομερά ενδιαφέρον και πρέπει να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν κάτι να πούνε, να μπορούν να μας εκπλήξουν, να μπορούν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Υπάρχει μια ισχυρή πίεση σήμερα στην τηλεοπτική αγορά να βγάζουμε πρόσωπα τα οποία να είναι επιθετικά να... και λειτουργεί και ο ανταγωνισμός ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός και απότομος. Πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε επίσης ε, και την άποψη που λέει ότι εμείς είμαστε το επίσημο κανάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και δεν μας βλέπει ο κόσμος τα σοβαρά. Αυτή είναι αντιλήψεις οι οποίες δύσκολα μπορεί να καταπολεμηθούν βέβαια. Έχουμε όμως ένα τεράστιο πλεονέκτημα, την πολυγλωσία. Πιστεύουμε ότι η πολυγλωσία είναι ένα τρομακτικό πλεονέκτημα του Euronews, πρέπει να συνεχίσουμε να το επιδιώκουμε και γι' αυτό παράγουμε και ευρωπαϊκές εκπομπές στις χώρες, στη γλώσσα τους. Δεν έχουμε χώρο και στη Λιόν, δεν μπορούμε να εργαστούμε με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο ρυθμό και να παράγουμε προϊόντα στη Λιόν σε πέντε γλώσσες ταυτόχρονα γιατί οι δημοσιογράφοι ναι μεν έχει ο καθένας τη γλώσσα του αλλά συνεργάζονται και στις υπόλοιπες. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να απευθυνθούμε στους λαούς σε τοπικό επίπεδο και δεύτερον αυτή η πολυγλωσία ταυτόχρονα δίνει και δυνατότητα για διαφορετικές θα έλεγα κρίσεις από αλόγλωσσους κάθε ξένος αν θέλετε δημοσιογράφος βλέπει την είδηση στη γλώσσα του και πηγαίνει και γράφει ξανά την είδηση στη γλώσσα του. Σαν παράδειγμα η ελληνική ομάδα για την ελληνική κρίση θα εξηγήσει στον γερμανό δημοσιογράφο τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κρίση αυτή και έτσι εμπλουτίζεται ο τρόπος λειτουργίας του γερμανικού τμήματος. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανάμιξη εμπειριών και πλούτου λόγω της χρήσης των πολλών γλωσσών. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Η τελευταία είναι να μιλήσουμε για την Ευρώπη των πολιτών. Είμαστε καλοί στην Ευρώπη φυσικά τη θεσμική, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και για την Ευρώπη των πολιτών. Ε, το Eurovision, τα λαχεία Euromillion, ή και το θέμα του έρασμου, το έρασμους για μένα επειδή με της γενιάς του έρασμου είναι κάτι το μαγικό. Υπάρχουν τέτοια ονόματα, λίγα θα έλεγα, τέτοια μπραντ για την Ευρώπη και πρέπει να τα προωθούμε, πρέπει έτσι να φτάσουμε στην Ευρώπη των πολιτών, στην Ευρώπη των Ευρωπαίων. Δύο επιπλέον παραδείγματα για να σας πω τον τρόπο με τον οποίο Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Ξέρετε ότι ανοίγουμε τα γραφεία μας στις Βρυξέλλες, ε, μπορείτε να τα επισκεφθείτε, είστε καλοδεχούμενοι. Ε, σε πέντε γλώσσες δουλεύουμε σε αυτά τα γραφεία και θα γιορτάσουμε και το πρώτο έτος λειτουργίας του γραφείου το Σεπτέμβριο. Και με την κυρία Ρέντινγκ θα είναι εκεί και θέλω να συναντηθούμε πάλι. Ένα άλλο παράδειγμα Ίσως ήμασταν το μόνο κανάλι στον κόσμο που γιορτάσαμε την ημέρα της Ευρώπης σε όλη την διάρκεια της ημέρας ασχοληθήκαμε με την Ευρώπη. Είχαμε και μία συνέντευξη του Πρόεδρου Βαν Ρόμποϊ. Ε, des, euh, des personnes qui euh, ο Βαρομπάη λοιπόν μπόρεσε να ακουστεί και φυσικά του τέθηκαν ερωτήσεις, διαδραστική εκπομπή και στις Ηνωμένε Πολιτείες και στη Βραζιλία και στην Τουρκία, εκτός Ευρώπης δηλαδή. Έχω πέντε λεπτά, αλλά δεν θα τα εξαντλήσω. Τα υπάρχουν ε, λοιπόν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ποιος τα χρηματοδοτεί και τι χρηματοδοτούν και αυτά με τη σειρά τους. Κατάρχας έχουμε ε, χρήματα από διάφορες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρηματοδοτούν ορισμένα προγράμματα που κρατάνε ένα χρόνο ή ένα μήνα. Ε, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Δικαιοσύνης, Εκπαίδευσης, Εξωτερικών Υποθέσεων Πρόκειται δηλαδή για επιμέρους προϋπολογισμούς οι οποίοι καλύπτουν το κόστος των εκπομπών, ειδικών εκπομπών. Και έχουμε και ένα γενικό ε, πλαίσιο συμφωνία με τη Γενική Διεύθυνση ε, Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες εκπομπών. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες αυτών των επιμέρους εκπομπών αλλά νομίζω τις ομάδες των εκπομπών. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε πολλές εκπομπές που έχουν τόσα προγράμματα για την Ευρώπη. Το iTalk σαν παράδειγμα, το UTalk για τον πολίτη, το Ευρωπαϊκό Network που υπάρχουν τρεις συζητητές Ταυτόχρονα Έχουμε το Europe Weekly κάθε την εβδομάδα που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά θέματα απευθείας από το γραφείο. Έχουμε το Close Up Europe Έχουμε γενικά τους ρεπόρτες, ένα, μια εκπομπή θα έλεγα για μεγάλα ε, ρεπορτάζ. Έχουμε επίσης το SMS Planet για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Generation Y ε, για την γενιά Y λέει ο μιλητής, ε, το Metropolitans που αναφέρεται στην προβληματική του κέντρου των πόλεων, το EU Crime που ασχολείται με τα θέματα τα ποινικά και του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, από το 2013 θα έχουμε εκπομπή για τα, ευρωπαϊκά, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τη μετανάστευση και για το διάστημα πάρα πολύ σύντομα. Στο τέλος θα σας δείξω έναν πίνακα για να προσπαθήσω να σας πείσω, δεν ξέρω αν σας έπεισα, αλλά προσπαθήσαμε είναι ένας πίνακας ο οποίος συγκρίνει το Euronews με το France 24, το Deutsche Welle, το Al Jazeera και το, ε, Russian, ε, το ρωσικό κανάλι ενημέρωσης. Βλέπετε εδώ τις επιδόσεις ε, του Euronews σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Εμείς παίρνουμε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο, 20% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από τις επιμέρους δημόσιες υπηρεσίες, τα δημόσια κανάλια, τα κρατικά κανάλια κάθε χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Φίλιπ Κέλλαρ που είναι εδώ που έχει προετοιμάσει τον πίνακα. Ενώ βλέπετε λοιπόν ότι το κόστος των άλλων καναλιών είναι 100 εκατομμύρια για το France 24, 100 για την Deutsche Welle και τα και Al Jazeera 100 και Russian News 65 αυτοί δουλεύουν σε μία ή σε δύο γλώσσες το καθένα από αυτά τα κανάλια. Ενώ εμείς με τα χρήματα αυτά τα λιγότερα δουλεύουμε σε πέντε καταρχάς γλώσσες και σε πολύ περισσότερες μετά. Βλέπετε λοιπόν ότι το κόστος, η σχέση κόστους και επίδοσης είναι ε, πάρα πολύ ε, καλύτερη σε εμά από ό,τι στο Αλτζαζίρα. Επίσης η διείσδυσή μας στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Βλέπετε ότι έχουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις από ότι οι ανταγωνιστές μας. Έχουμε 31% εμείς, ενώ οι άλλοι δεν ξεπερνούν το 5 ή το 10%. Βλέπετε ότι σε σχέση με το κόστος των 6 λεπτών που επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να μπούμε σε τόσα πολλά νοικοκυριά, ενώ σε ανταγωνιστικά κανάλια το αντίστοιχο κόστος είναι πάνω από 1 ευρώ. Εμείς εδώ συσχετίζουμε αν θέλετε ε, το, τα χρήματα που επενδύουμε σε σχέση με τον αριθμό αυτών που βλέπουν το κανάλι. Βλέπετε ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια πάλι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι ένα προς τρία. Οι αριθμοί ομιλούν από μόνοι τους και αντιπροσωπεύουν θα έλεγα ένα καλό κλείσιμο αυτής της παρουσίασης σχετικά με την αποτελεσματικότητα λειτουργίας και τη σωστή χρήση των ποσών των κοινοτικών από τη Euronews. Όπως έλεγε ένας Γάλλος πολιτικός, βοηθήστε με, δηλαδή βοηθήστε μας. Ήσασταν αρκετά πιστικός. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Λόκεγκάρτ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας δείξατε πολλά αριθμητικά στοιχεία, αλλά και πολύ πιστικά επίσης. Ε, θέλω να σας, ε, να σας συγχαρώ λοιπόν για τις προσπάθειές σας. Τα πάτε πολύ καλά. Είστε ένα ζωντανό παράδοξο νομίζω. Δημιουργηθήκατε σαν το πρώτο πανευρωπαϊκό μέσο ε, και κατά τη γνώμη μου παραμένετε το μόνο. Αυτό λέει πολλά και για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε. Νομίζω ότι πολλά πράγματα συνέβησαν στον κόσμο και στον κόσμο των μίδια από τότε που αρχίσατε εσείς. Έχουμε μια πολύ κατακαιρματισμένη εικόνα ε, σήμερα. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αναμφίβολα έχετε επιτύχει κάτι μπορείτε να ε, προσεγγίσετε πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη. Ε, πολλοί σας παρακολουθούν, αλλά στη Δανία, που είναι η χώρα μου, πρέπει να σας πω ότι κανένας Δανός δεν κοιτάζει το Euronews. Μετά από 20 χρόνια, λοιπόν, φαίνεται ότι κάποιες περιοχές της Ευρώπης δεν τις έχετε καλύψει. Δεν τις έχετε πλησιάσει. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για σας. Αν θέλετε την υποστήριξη όλων των Ευρωπαίων, αν μιλάμε για χρήματα και για οικονομική υποστήριξη. Νομίζω. Μια καλή ερώτηση λοιπόν είναι ποια είναι η φιλοδοξία σας, τι θέλετε να γίνετε. Εγώ έχω κάποιες ιδέες γιατί έχω συνομιλήσει μαζί σας και έχω επισκεφθεί και τα γραφεία σας ε, στις Βρυξέλλες. Συγχαρητήρια και για αυτά και σε λίγες μέρες θα πάω και στη Λιόν. Αλλά έχω ακόμα κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το ποια είναι η πραγματική σας φιλοδοξία. Θέλετε να ε, γίνετε το δημόσιο κανάλι της Ευρώπης. Και τι σημαίνει αυτό. Και αν αυτή είναι η φιλοδοξία σας, για πράγμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για 18 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο νομίζω. Γιατί αν θέλετε να επιτύχετε αυτό το στόχο, μιλάμε για πολύ περισσότερα χρήματα πιστεύω. Γιατί η παραγωγή στη τηλεόραση είναι ακριβή. Και αυτό είναι από τα προβλήματα βέβαια. Ε, παρακαλώ λοιπόν να είστε ειλικρινείς ε, απέναντί μας και να μας πείτε αν αυτή είναι η φιλοδοξία σας και αν όντω είναι, πώς μπορούμε να την ε, ε, επιτύχουμε από κοινού και τι ε, χρήματα θα χρειαστούν, ώστε να κάνουμε τη σχετική συζήτηση κατά τα επόμενα χρόνια και να ανακαλύψουμε τι πρέπει να γίνει. Και κάτι που με ανησυχεί λιγάκι. Λέτε ότι μπορείτε να προσεγγίσετε τόσους ανθρώπους και μία από τις προκλήσεις είναι να πιάσετε τις ελίτ. Μάλλον τις ελίτ είναι, οι είναι οι ομάδες που μπορείτε να πιάσετε τώρα. Και υπάρχουν και οι άλλοι. Ε, μιλάμε για ε, ότι έχετε αυτή τη στιγμή ε, πρόσβαση σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους και θέλετε να έχετε σε 350 εκατομμύρια. Λείπουν δηλαδή 345 ε, εκατομμύρια. μπορείτε να το κάνετε. Γιατί αν δείτε τα νούμερα του CNN και άλλων, ε, βλέπετε ότι εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομάδες του κοινού για να είναι leaders σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της αγοράς. Ε, φιλοδοξία σας λοιπόν, το, ο σκοπός σας είναι να πιάσετε το ευρύτερο κοινό, να έχετε περιφερειακά και τοπικά νέα ή να είστε στην πλατφόρμα που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, να είστε οι ειδικοί των νέων από τις Βρυξέλλες, των νέων από την Ουάσιγκτον. Θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας επ' αυτού, γιατί δεν νομίζω ότι μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να ε, κάνετε και τα δύο πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στρατηγική σημασία πιστεύω και θα ήθελα τα σχόλιά σας επ' αυτού. Ίσως θα μπορούσα να επανέλθω και για άλλα θέματα. Ε, ο συνάδελφος πάντα με τη στρατηγική ασχολείται. Μπορείς και μετά Χέλγκα Τρίπελ. Um, ε, θα μαζέψουμε τι ερωτήσει και θα απαντήσετε. Σα ευχαριστώ. Πρώτο ερώτημα. Νομίζω πως με παρεξηγήσατε. Ρώτησα το εάν το πρόγραμμα Media θα συνεχιστεί. Αλλά εγώ το σήμα, για το σήμα ρωτούσα. Το λογότυπο γιατί μου, μας είπε η κυρία Επίτροπος θα φύγουν όλα τα σηματάκια. Όλα τα λογότυπα. Εν πάση περιπτώσει. Βεβαίω όλοι θέλουμε ε, αξιόπιστες ε, πληροφορίες για το τι αποφάσεις λαμβάνονται στην Ευρώπη. Όλοι οι λαοί σήμερα έχουν προβλήματα με το υψηλό κόστος των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Και καμιά φορά οι ειδήσει για τα ευρωπαϊκά είναι μόνο σκάνδαλα. Το ερώτημά μου λοιπόν. Μήπως καλύτερη χρήση θα ήταν να επικεντρωθούμε σε ένα βασικό σταθμό και όλοι οι υπόλοιποι, πολωνικά και τα λοιπά, να μεταδίδουν το ίδιο πρόγραμμα απλά, σε άλλη γλώσσα. Γιατί ξέρω πως το κόστος παραγωγής είναι το μεγάλο Γι' αυτό ακριβώς ε, δεν ε, υπάρχουν ανταποκρίσεις για τα ευρωπαϊκά. Και άρα θα έπρεπε εσείς να κάνετε παραγωγή εκπομπών οι οποίες μετά θα μεταδίδονται από τους υπόλοιπους. Κυρία Τρούπελ, ευχαριστώ τόρς. Όταν κατάλαβα αυτά τα οποία μας εξηγήσατε, η ιδιαιτερότητα του Euronews είναι πως ε, μέσα στη μεθοδοργασία σας έχετε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν από ολόκληρη την Ευρώπη και μεταφράζουν στη γλώσσα τους και πραγματικά παράγουν ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι σχετικό με αυτό το οποίο είπε άλλος Εάν μπορούσατε να μας πείτε το ποιο θα είναι το μέλλον το οποίο θα επιθυμούσατε για τον κοινωνίο, ποια θα ήταν η απάντηση δεδομένης της κρίσης και τις ε, αρχές συνομιλίας για μια οικονομική και νομισματική ένωση. Εάν πετύχαινε κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν κρίσιμη σημασία να επεκταθεί το Euronews πολύ περισσότερο για να καλύπτει ε, αυτό τον ευρωπαϊκό χώρο Γιατί βεβαίω είναι κατακαιρματισμένη η κάλυψη, δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Αν όμω πάμε προ μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δεν θα έχει κάποιο αντίκτυπο αυτό στι ανάγκε και στην αναγκαιότητα του κύριου Καμία άλλη ερώτηση. Έχετε το λόγο. Έχω συνηθίσει σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Είναι οι ερωτήσεις που μας θέτουν οι μέτοχοί μας πρόσφατα για τη μελλοντική στρατηγική του Euronews που μας ζητούν να διευκρινίσουμε ποιες είναι ακριβώς οι φιλοδοξίες μας για τα επόμενα χρόνια. Συμφωνώ μαζί σας λέγοντας ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση, σε ένα ενδιάμεσο θα έλεγα χρόνο. Έχουμε πετύχει αρκετούς στόχους, ορισμένους στόχους, αλλά η η στόχη αυτή, η επίτευξή τους θέτει ερωτηματικά για τις μελλοντικές εξελίξεις. Έχουμε εργαστεί λοιπόν σε ένα νέο στρατηγικό πρόγραμμα 12-14 που παρουσιάστηκε και στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας αμέσως μετά την παρουσίαση της ε, πρότασης αυτής στους μετόχους. Θα σας το παρουσιάσουμε όταν έλθετε στη Λιόν. Υπάρχουν δύο βασικοί άξονες. Καταρχάς, στόχος του Νιούρνιους είναι En fait, euh, que nous sommes peut-être euh, Θέλουμε να γίνουμε ένα μέσο το οποίο να σας εξηγήσω τι θέλουμε να πούμε ακριβώς. Να έχουμε τοπική αλλά και διεθνή διάσταση ταυτόχρονα. Δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τους ανταγωνιστές μας, οι οποίοι θα έλεγα έχουν κάποιες μονομερείς τάσεις δηλαδή όπως η Deutsche Welle, η France 24, μια εθνική, αν θέλετε, διάσταση, καθοριστική, η Al Jazeera μια πολιτιστική, αλλά ε, μονομερή ελαφρώς. Ενώ εμείς στην ουσία είμαστε ο ΙΕ της τηλεόρασης, είμαστε το μοναδικό κανάλι το οποίο έχει στην αίθουσα σύνταξης πάρα πολλά και διαφορετικά προϊόντα. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ γιατί ίσως κατάλαβα λάθος την κυρία Τρούπελ. Δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα εγώ τι ακριβώς είπατε μέσω της μετάφρασης. Το 99% του κόσμου θεωρεί ότι το News» ε, γράφεται και γυρίζεται σε μία γλώσσα και μεταφράζεται σε 10 άλλες. Έτσι πίστευε ο κόσμος παλιά, ότι οι διάφορες γλωσσικές εκδόσεις του Euronews είναι μεταφράσεις. Δεν ισχύει αυτό βέβαια. Οι διαφορετικές γλωσσικές μορφές του Euronews δεν είναι μεταφράσεις, είναι script, πρωτότυπες, γραμμένα από τους δημοσιογράφους της κάθε σύνταξης και το βίντεο ναι μεν είναι το ίδιο αλλά αυτό που ακούμε, το ακουστικό κομμάτι διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα και αυτό αν θέλετε δικαιολογεί ε, το κόστος ε, ε, της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν χρηματοδοτεί την μετάφραση αλλά πραγματικά εθνικά επιμέρους σχόλια. Σήμερα λοιπόν το Euronews είναι ανάμεσα σε ένα τοπικό ας πούμε ε, κανάλι, εθνικό κανάλι ενημέρωσης και σε, κάποιες, ε, ε, σε κάποια κανάλια έτσι, διεθνή αλλά και μονομερή όπως με το, το CNN και τα λοιπά. Προσπαθούμε να είμαστε λοιπόν να είμαστε σφαιρικό κανάλι αλλά με τοπικές ε, νότες, με τοπικές αποχρώσεις. Δηλαδή δείχνουμε διαφορετικού τύπου βίντεο γιατί σε εμά αυτό το μοναδικό βίντεο που δείχνουμε στις διάφορες γλώσσες είναι ένα πρόβλημα γιατί τεχνικά μας αναγκάζει να μιλήσουμε περίπου με τον ίδιο τρόπο στους Αμερικανούς, τους Ασιάτες και στους Ευρωπαίους έχουμε περίπου το ίδιο περιεχόμενο, ενώ η ιδέα που πιστεύουμε ότι είναι σωστή και τη συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ιδέα πολύ φιλόδοξη και ανταποκρίνεται, αν θέλετε, και σε επίπεδο φιλόδοξων πόρων, θα είναι σε μια πρώτη φάση να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο Euronews κόσμος και στο Euronews Ευρώπη, δύο διαφορετικές ταυτότητες οι οποίες θα είναι κατά 90 ή 95% όμοιες, το περιεχόμενο δηλαδή ε, του Euronews κόσμος θα είναι ίδιο κατά 90% ή 95% με το Euronews Ευρώπη, αλλά το 5% θα διαφέρει για τον υπόλοιπο κόσμο, θα είναι καταλληλότερο ή για την Ευρώπη. Έτσι θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις αγορές μας πολύ περισσότερο γιατί σήμερα δυσκολευόμαστε να πείσουμε τους Ασιάτες το Εράσμο σαν παράδειγμα άμα πείτε ε, εσείς μιλήσετε για το Εράσμο στο Χονγκ Κονγκ ε, είναι πεπισμένοι ότι ασχολείστε μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, εμείς μιλάμε για τον κόσμο, για όλο τον κόσμο, αλλά με, μια, με ένα όραμα ευρωπαϊκό, με μια αντίληψη ευρωπαϊκή. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε περισσότερο τις αγορές αυτές, να μπούμε περισσότερο στις αγορές, ε, πιο συγκεκριμένα πάνω σε ένα, σε ένα δεκάλεπτο δελτίο ειδήσεων, σαν παράδειγμα που περιλαμβάνει 10 θέματα, ένα-ενάμιση λεπτό το καθένα, να περιλαμβάνει ένα επιπλέον τοπικό θέμα σε σχέση με το ευρωπαϊκό και να ταξινομούμε διαφορετικά τα θέματα διαφορετικά αν είστε στην Ευρώπη, στην Ασία ή ε, στην Αμερική. Γιατί το τρίτο θέμα σε ένα δελτίο ειδήσεων δεν ε, έχει την ίδια ιεράρχηση σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε και πιο διεισδυτικοί στις αγορές. Πρέπει ακριβώς να κερδίσουμε την επιρροή μας μέσω της πολυγλωσσίας και της παρουσίας μας στις αγορές. Η ελληνική περίπτωση είναι πολύ συγκεκριμένο, αν θέλετε, παράδειγμα, προσπαθούμε να παράγουμε επιτόπου. Ε, στην, στην Ελλάδα λειτουργούμε με ψηφιακό δίκτυο επίγειο. Και δεν ξέρω, από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει στην Ελλάδα στα ελληνικά ενημερωτικό κανάλι που να μεταδίδει μόνο ειδήσει. Λοιπόν, αν εμείς μπορέσουμε με τοπικό τρόπο σε κάθε γλώσσα να παράγουμε τις ειδήσει που ενδιαφέρουν τοπικά, πρώτον θα μειώσουμε το κόστος και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Πάκα αναφέρθηκε προηγουμένως σε ένα προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα 7 εκατομμύρια σήμερα χρηματοδοτούν και τα ελληνικά, την ελληνική υπηρεσία, την ουγγρική υπηρεσία και την πορτογαλική υπηρεσία. Δηλαδή για το κόστος μίας γλώσσας, ας πούμε στα φαρσί ή στα αραβικά γύρω στα 5 εκατομμύρια εδώ και 5 χρόνια. Τώρα με τα ίδια λεφτά καλύπτουμε τρεις γλώσσες και το κόστος τριών γλωσσών γιατί έχουμε την παραγωγή επιτόπου, ξέρετε ότι στη Γαλλία το κόστος των μισθών είναι υψηλότερο, η κοινωνική πρόνοια κοστίζει περισσότερο, το κόστος εργασίας είναι υψηλό ενώ στις άλλες χώρες μπορεί να είναι χαμηλότερο. Δεύτερον, όταν είμαστε επιτόπου παρόντες ε, μπορούμε να είμαστε πιο διεισδυτικοί, να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή στις τοπικές αγορές. Θα έχουμε 30 δημοσιογράφους στην Αθήνα, 30 στην ε, Βουδαπέστη, τοπικούς ανταποκριτές και θα μπορούμε να είμαστε και πιο αναγνωρίσιμοι από τον τοπικό πληθυσμό. Σε σχέση με το CNN εμείς πιστεύουμε ότι αν το κάνουμε αυτό τότε μαθηματικά αν θέλετε, αριθμητικά θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες με αυτήν την υπηρεσία που θα παράγουμε στην Ελλάδα από Έλληνες παραγωγούς, περισσότερες δυνατότητες να μας δούνε περισσότεροι θεατές στην Ελλάδα. Το CNN δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Η βασική ιδέα είναι λοιπόν να ανοιχτούμε σε 20, σε 30 γλώσσες με αυτό το σύστημα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν στη Λιόν. Μπορούμε λοιπόν να καλύψουμε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τελευταίο σημείο. Έχουμε ένα πρόβλημα που είναι το ψηφιακή επίγεια τηλεόραση. Είναι ένα θέμα... Et, ε, ε, il y a donc de nouveaux entrants. Η επίγεια λοιπόν ψηφιακή τηλεόραση σε κάποιες χώρες ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και περνάμε από δορυφορικά μέσα και πληρώνουμε το κόστος. Και αυτό μπορεί να κοστίζει 15 εκατομμύρια στη Γαλλία, 2 εκατομμύρια στην Ελλάδα ή στην Πορτογαλία. Πολύ ψηλό το κόστος. Και εδώ έχουμε πρόβλημα γιατί η σχόρησή μας δεν είναι ικανοποιητική. Υπάρχουν πάρα πολλά τοπικά κανάλια που είναι παρόντα σε ψηφιακό επίγειο τρόπο μετάδοσης. Ο προϋπολογισμός μας λοιπόν που θα μας επέτρεπε να είμαστε παρόντες σαν ε, δημόσια ευρωπαϊκή αν θέλετε τηλεόραση θα έχει θετικά αποτελέσματα νομίζω συνολικά για μας. Συμπερασματικά λοιπόν η βασική ιδέα είναι να μην γίνουμε ένα μαζικό κανάλι mass media, αλλά να πούμε ότι έχουμε δύο στόχους. Πρώτον, να είμαστε παρόντες σε όλο τον κόσμο. Ε, δεν μπορείτε να φανταστείτε σε ποιο βαθμό είμαστε δημοφιλείς στη Ρωσία σαν παράδειγμα η Ρωσία είναι ο μισός, οι μισοί θεατές του Euronews είναι στη Ρωσία, στην κεντρική Ευρώπη, στην Αστάνα, στον Πακού. Τρελαίνονται για την Ευρώπη και βλέπουν το Euronews. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να μείνουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό διεθνές επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε ένα στόχο ευρωπαϊκό όχι για να φτάσουμε όλο τον ευρωπαϊκό πληθυσμό και να τον καλύψουμε, αλλά να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων. Και γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να αναγνωριστούμε σαν ένα κανάλι κοντά στον Ευρωπαίο. Είμαστε αναγνωρισμένοι σαν ευρωπαϊκό θεσμικό κανάλι. Βασικός μας στόχος είναι αυτός και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε. Αλλά θα το συμπληρώσουμε αυτό όντας κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη. Σαν παράδειγμα, να, να δείχνουμε τα αποτελέσματα του Euromillion, να δείχνουμε τη στοιχεία του έρασμου, ταξίδια ευρωπαϊκά. θα δημιουργήσουμε ας πούμε και το Euronews Talents, το οποίο θα επιτρέπει να αναζητούνται ε, ταλέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε δύο πρότυπα, το ένα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο θα απονείμουμε στις Βρυξέλλες και θα ζητήσουμε από τις εταιρείε να συμμετέχουν. Κάνουμε επίσης ένα μεγάλο μουσικό διαγωνισμό με συγκροτήματα στην Ευρώπη. Τα συγκροτήματα θα μας στείλουν μακέτες και θα επιλέξουμε. Και τέλος, προσπαθούμε λοιπόν να μην χάσουμε την θεσμική διάσταση. Έχουμε μια μεγάλη τύχη που συνεργαζόμαστε μαζί σας γιατί εμείς θεωρούμε ότι εσείς σαν θεσμικό όργανο είσαστε ο πρώτος μας πελάτης. Σας βλέπουμε σαν πελάτη, αυτό είναι κανονικό και σας σεβόμαστε σαν πελάτη. Έχουμε μεγάλη τύχη λοιπόν, γιατί σε σχέση με όλες τις κριτικές που υφιστάμεθα, να πω ότι ποτέ, ποτέ δεν μας πίεσε κανείς σε επίπεδο συντακτικό από πλευράς του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, Έχουμε μια όριμη σχέση, έχουμε ανθρώπους απέναντί μας οι οποίοι μας εμπιστεύονται, μας δίδουν χρήματα και μας βοηθούν να κάνουμε τη δουλειά μας με ανεξάρτητο τρόπο. Ευχαριστώ για το τελευταίο σας συμπέρασμα. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Το συζητήσαμε σήμερα και σε αυτό. Δεν πρέπει να ασκούμε πιέσει και δεν ασκούμε. Και ευχαριστώ που το διαπιστώσατε. Χαίρομαι που απαντήσατε τόσο αναλυτικά και ο κύριος Λόκεγκαρτ νομίζω ικανοποιήθηκε με τις στρατηγικές του σκέψεις. Σας ευχόμαστε, μα, αν βλέπω τους συναδέλφους νομίζω πως συμφωνούν. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στο νέο σας αυτό εγχείρημα που είναι ευρωπαϊκό αλλά και προσανατολισμένο προς τον κόσμο και ελπίζω να έχουμε λεφτά να σας στηρίξουμε αλλά πρέπει να τα πάρουμε για να τα δώσουμε τα λεφτά έτσι. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε στη... οι κυβερνήσεις να πιστούν και αυτές για τη δουλειά που κάνετε εμείς. Ε, πάντως είμαστε πεπισμένοι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τι ήτανε? Α, τίποτα μάλιστα. Είμαι ναι, ε, Μάλιστα, 16. Συνάντηση των συντονιστών έγινε το μεσημέρι. Διάφορα. Θέτε τίποτα για τα πρακτικά. Όχι. Εγκρίνονται διάφορα. Τίποτα τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διερμηνείς. Καλώς σας βράδυ.